Καλώ ήρθατε λοιπόν όλε και όλοι. Θα ήθελα να χαιρετήσω την αντιπροσωπεία γεωργών από την Αυστρία, την Καρινθία. Καλώς ήρθατε. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα Ιουλίου θα πάμε στην Αυστρία και θα γνωρίσουμε, θα τα ξαναπούμε και στην πατρίδα σας. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 23ης και 24ης Ιανουαρίου. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις, πριν το τέλος της συνεδρίασης θα εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών. Σημείο 3. Ανακοινώσει του Προέδρου. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι, όπω ξέρετε, το 2012 είναι το έτο τη 50 η επαιτίου τη ε, κοινή αγροτική πολιτική τη ΚΑΠ. Για να γιορτάσουμε αυτή την επέτειο, θα ήθελα να σα προσκαλέσω όλου σε μία δεξίωση που θα κάνουμε εδώ, στο Κοινοβούλιο, στι 19 Μαρτίου, στις 7.30 ώρα το απόγευμα έχω προσκαλέσει σε συνεργασία με την Δανέζικη Προεδρία και τους Υπουργούς Γεωργίας όλων των κρατών μελών. Και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να συναντηθούμε και να έχουμε και άτυπες επαφές για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Στις 19 λοιπόν Μαρτίου, στις 7.30 το απόγευμα, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια της ΚΑΠ. Μαζί με το Συμβούλιο Γεωργίας, τους Υπουργούς δηλαδή Γεωργίας. Πολύ ωραία. Αν είστε έτοιμοι, πάμε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης. Έχετε όλη την κάρτα ψηφοφορία σας, ελπίζω, άχρια να ψηφίσουμε. Μιλάμε για την ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοπικιλότητα. Η συγγητής είναι η Βασίλικα Βιόρικα Νταντσίλα. Έχει ετοιμάσει μία γνωμοδότηση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοπικιλότητα μέχρι το 2020. Παρουσιάστηκαν 59 τροπολογίες. Η γνωμοδότηση θα πάει στην έκθεση για να εξεταστεί στην έκθεση που ετοιμάζει η Επιτροπή ΕΝΔΗ, η Επιτροπή Περιβάλλοντο, η οποία είναι καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Η ψηφοφορία στην ΕΝΔΗ θα γίνει στι 29 Φεβρουαρίου. Ο κατάλογο ψηφοφορία είναι και αυτό προσαρτημένο ε, στο κείμενό σα και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε τις ε, ψηφοφορίες. Είσαστε όλοι, λοιπόν. Ξεκινάμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 2-1. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήσατε όλοι. Δεν δουλεύει το μηχανημά σας. Ψηφίζουμε ακόμα, ψηφίζουμε, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Έχουμε μία ψήφο επιπλέον του ΕΛΚ, μία παραπανήσια ψήφο του ΕΛΚ. Έχουμε κλείσει το μεταξύ τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε στην παράγραφο 2.2. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται νομίζω. Σωστό. Απορρίπτεται. Τροπολογία νούμερο 1. Πόλσεν. Ψηφίζουμε. Ένα ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τρίτη τροπολογία. Ψηφίζουμε. Άλβες. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τέταρτη τροπολογία. Πάξας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται νομίζω. Σωστό. Ψηφίζουμε την πέμπτη τροπολογία Σιλβέστρης. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται νομίζω. Ναι. Αριθμός 6. Μποβέ και λυπή. Πέρας. Απορρίπτεται. ψηφίσουμε την παράγραφο 2, τροπολογία 7. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 8. Καλινόφσκι. Ψηφίζουμε ακόμα. Πέρας. Εγκρίνεται. 13. Γιάρ και άλλοι. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έχουμε μία ψήφο παραπάνω από το ΕΛΚΑ. Ελέγξτε παρακαλώ τις ψήφους σας. Ψηφίζουμε. Τη 14. Πέρας. Απορρίπτεται. 16. Πόλσεν. Διορθώνει ο πρόεδρος. Τη 15 πρώτα. Νταντά. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 τώρα. Πόλσον. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη. Όταν κάνουμε μια ψηφοφορία ηλεκτρονική, πρέπει να βλέπουμε το αποτέλεσμα και να βλέπουμε το σχετισμό δυνάμεων. Δεν εμφανίζεται όμω. Κρίμα δεν είναι. Δεν μπορούν οι τεχνικοί να μα επιτρέψουν να βλέπουμε το αποτέλεσμα τόσο ώστε να βλέπουμε ποιοι ψηφίζουν, ποιοι καταψηφίζουν. Μερικέ φορέ είναι ενδιαφέρον το βλέπουμε. Λοιπόν, είναι διαφωτιστικό. Ναι, Μάρκ. Θα προσπαθήσουμε να σα δείχνουμε στι οθόνε τα αποτελέσματα. Μπορείτε να δώσετε κατάλληλε οδηγίε. Εμεί συνεχίζουμε στο μεταξύ. Εγκρίναμε την ε, τροπολογία 16 και τώρα ψηφίζουμε τη 17. Σικεριέσκη. Πέρας. Εγκρίνεται νομίζω. 22 υπέρ, 15 κατά. Καμία αποχή. 18. 18. Ψηφίζουμε τη 18. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσουμε τη 18. Εγκρίνεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 35 ψηφι... υπέρ, 2 κατά. 19. Ψηφίζουμε τώρα τη 19. Πέρας ψηφοφορίας. Η 25 ψηφιπέρ υπέρ, 10 ψήφι κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 20. Σάρμπο. Ψηφίζουμε την τροπολογία του Σάρμπου. Πέρας της ψηφοφορία τη τροπολογίας 20 εγκρίνεται με ευρεία πλειοψηφία. 31 ψήφι υπέρ, 6 ε, κατά. 21. Νεντελτσέβα. Ψηφίζουμε τώρα. Μαρία, σας πένσε εδώ, ε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24 ψήφι υπέρ και 13 κατά. 22. Ψηφίζουμε τώρα την 22. Πέρας. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 32 κατά, 4 υπέρ απορρίπτεται. 23. Τελάνζο. Πέρα στις, 20, τις ψηφοφορίες για την 23, αποτέλεσμα, 26 ψήφοι υπέρ, 10 κατά, εγκρίνεται βέβαια. 24. Όχι, έχει αποσυρθεί. 25. Ψηφίζουμε την 25 και στην ΚΕΡ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27 ψηφιπέρ. 10 κατά. Λυπάμαι, Μάρκ, το σύστημα δεν λειτουργεί, οπότε πρέπει να επαναλαμβάνω εγώ τα νούμερα. 26. Ψηφίζουμε την 26. Γιάρ και Λυπή. Πέρας προφορίας. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Μεγάλη πλειοψηφία. 32 ψήφοι υπέρ, 4 κατά. Τώρα λειτουργεί. Πολύ ωραία. Λειτουργεί και το σύστημα. Ψηφίζουμε την 27. Πέρας προφορίας. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Εγκρίνεται πάντως. 28. Ψηφίζουμε την 28. Πέρας. 28 απορρίπτεται με 33 ψήφους κατά, 4 υπέρ. 29. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται νομίζω. Με 36 ψήφους κατά. 30. Λαδία. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Συγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 32. Ψηφίζουμε 32. Πέρας ψηφοφορίας, 32, η 32 εγκρίνεται με 20 ψηφούς υπέρ, 18 κατά. 33. Πέρας. Απορρίπτεται. 34. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε 36. Ταραμπέλα. Ψηφίζουμε την 36. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η τροπολογία αυτή ...είναι μεγάλη πλειοψηφία. Μία ψήφο κατά μόνο πήρε. 37. Πέρας προφορίας. Απορρίπτεται. Τριανταοχτώ. Πέρα ψηφοφορίας. εκκρίνεται νομίζω, όντως. Με 25 ψήφους υπέρ και 11 κατά. Τώρα ψηφίζουμε την 39. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία. 40. Ταραμπέλα. Ψηφίστε τώρα. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Και αυτή. Και τώρα τη 41. Ταραμπέλα πάντα. Πέρας. Απορρίπτεται. 42. Ντόρφμαν. Τέλος της ψηφοφορίας. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Όντως. 49. Ταραμπέλα. Πάλι. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ψηφίζουμε την 50. Τέλος. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 52. Ταραμπέλα πάλι. Ψηφίζουμε την 52. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 53. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 54. Πόλσεν και άλλοι. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 55. Παράγραφος 6. Σάρμπου. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 56. Τανσίλα. Τέλος ψηφοφορίας Εγκρίνεται. 57. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 58. Νταντά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελευταία τροπολογία. Η 59 ταραμπέλα. Ψηφίζουμε τώρα. Την 59. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τελική ψήφος της νομοδότησης όπως την τροποποίησαμε. Ψηφίζουμε το συνολικό κείμενο, το τροποποιημένο. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, κυρία Νταντσίλα. Και τώρα. Πάμε στο εργαστήρι μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ξεκινάει τώρα το εργαστήριο για την αγροτική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή της νέας ΚΑΠ. Έχουμε ετοιμάσει πέντε εργαστήρια, ε, είναι το πρώτο από τα πέντε, και θα δούμε ειδικά θέματα της μελλοντική γεωργικής πολιτικής. Αυτά τα εργαστήρια μας ε, βοηθούν να ετοιμάσουμε τις εκθέσεις και τις τροπολογίες για τις νομοθετικές προτάσεις που μας έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Βάντεν Πλεκ από το Πανεπιστήμιο Βαγγενίκε που θα μας παρουσιάσει την, το κείμενό του και μετά θα δώσω το λόγο στους βουλευτές για σχόλια κτλ. Ευχαριστώ τον καθηγητή Βάντερ Πλούγκ και θα ακούσουμε την παρουσίασή του. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Κομισιόν που είναι και αυτοί παρόντες. Ε, Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ συμπαθητικά σας λόγια, κύριε Πρόεδρε. Ε, με μεγάλη χαρά ήρθα εδώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτό το εργαστήριο. Έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω και τις έχω οργανώσει σε τρεις ομάδες. Πρώτον, ποια είναι τα θετικά σημεία της νέας πρότασης για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Δεύτερον, ποια είναι τα αρνητικά σημεία ε, που εντοπίζονται οι κίνδυνοι. Και τρίτον, θα παρουσιάσω κάποια στοιχεία που είναι θετικά αλλά μπορούν να βελτιωθούν έτσι Και αυτά τα θέματα θα τα αναλύσω όχι μόνο επί τη βάση του κειμένου που έχω διανύμει και του κειμένου που έχουμε μάλλον, αλλά θα κάνω και συχνές αναφορές στην ε, αγροτική δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Η ανάπτυξη της υπαίθρου δεν είναι μια πολιτική. Είναι και κάτι το οποίο γίνεται στην πράξη. Είναι μια πρακτική που ακολουθούν πάρα πολλοί αγρότες σε όλη την Ευρώπη, αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν την αγροτική δραστηριότητα, προσαρμόζονται ε, στα καινούργια δεδομένα και έτσι έχουμε μια πολύ σημαντική μεταβατική διαδικασία. Η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου λοιπόν μπορεί να πετύχει μόνο εάν γίνεται με διαδραστικό τρόπο και σε στενή συνεργασία με τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται επιτόπου στη βάση της κοινωνικής πυραμίδας στην Ήπεθρο, στην εξοχή. Εξού και κάνω αυτή την αναφορά ε, στην κατάσταση που βιώνουμε στην πράξη στην Ευρώπη. Καταρχάς, το πρώτο το οποίο είναι σημαντικό Μιλούμε για τη συνέχιση της ε, πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου και αυτό είναι καλό και ειδικότερα ε, έτσι όπως έχουμε οι συνθήκες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή σχεδιάζουμε πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου με στόχο να ενισχύσουμε τις αγροτικές οικονομίες και να μπορέσει η Γεωργία να διαδραματίσει τον νέο ρόλο που της αναλογεί. Να βοηθήσει στην επάρκεια τροφίμων, στην ασφάλεια των τροφίμων ε, και να διατηρήσει τον πληθυσμό στις, ε, στην Ήπεθρο. Όλα αυτά όμως απειλούνται. Υπάρχει ο κίνδυνος των ε, καταρρεύσεων των αγορών σε ορισμένες περιοχές η αγροτική περιοχή επικεντρώνεται εκεί μόνο, ενώ άλλες αγροτικές οικονομίες τίθενται στο περιθώριο. Κάθε φορά που σημειώνονται πολύ μεγάλες ανισορροπίες μεταξύ της οικολογίας, της κοινωνίας και των αγορών, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να παρεμβαίνουμε πολιτικά, να ασκούμε πολιτική για να αποκαταστήσουμε τις ανισορροπίες. Και η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ανάληψης πολιτικών ευθυνών. Αυτό είναι μια πρώτη παρατήρηση. Κατά δεύτερο λόγο, δεν θα ε, έχουμε πια τους τέσσερις άξονες με την ακαμψία τους. Αυτό βέβαια περιλαμβάνει και κάποιους κινδύνους, ωστόσο ε, για να συνεχίσουμε να έχουμε υψηλό επίπεδο αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και για να συνεχίσουμε να έχουμε την προσέγγιση του leader θα πρέπει να ε, εξαλειφθεί αυτή η ακαμψία, επομένως η προσέγγιση μας είναι θετική. Ε, στις Τις προηγούμενες φορές απευθυνόμασταν στον αγρότη κάθε έναν ξεχωριστά, ο οποίος ήταν ένας παθητικός, παθητικός δέκτης, αν θέλετε, αποδέκτης των ωφελιών της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Τώρα σημειώνονται μια πολύ σημαντική αλλαγή. Μιλούμε για εταιρικέ σχέσεις, για δίκτυα, για ομάδες ε, συνεταιρισμούς αγροτών, ομάδες παραγωγών ε, οι ομάδες παραγωγών αναδύονται πλέον στο προσκήνιο ως ένας νέος ε, συνομιλητής. Και όλα αυτά θα γίνουν όλο και πιο παρόντα την επόμενη επταετία. Το πρασίνισμα του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι καν πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να έχουμε έξυπνους συνδυασμούς. Στον πυλώνα 1 το πρασίνισμα σημαίνει ότι όλοι πρέπει να κάνουν μικρά βήματα και στον πυλώνα 2 σημαίνει αυτό ότι και εκεί πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα. Συνδυάζονται οι δύο αυτοί οι μηχανισμοί και ο συνδυασμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα. Για να δούμε τώρα ε, τι αποτελεί πρόβλημα σε αυτή τη νέα πρόταση για την πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Είμαστε τώρα στην τρίτη επταετία πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου και πάντοτε οι στόχοι ε, χαρακτηρίζονταν από συνέχεια. Μιλούμε για την αηφορία, για την καταπολέμηση των προβλημάτων από την κλιματολογική αλλαγή, για την εδαφική συνοχή, μεταξύ άλλων από την πρώτη διατύπωση της υφιστάμενης πρότασης μέχρι και τη σημερινή πρόταση έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή έχουν προσθεθεί διάφορες προτεραιότητες που δεν υπήρχαν. Έξι προτεραιότητες συγκεκριμένα. Και κατά την άποψή μου οι προτεραιότητες αυτές οδηγούν σε έναν κάπως ολισθηρό δρόμο. Ελοχεύει ο κίνδυνος ε, να αλλάξει το σημείο εστίασης, το σημείο στο οποίο δίνουμε έμφαση στην πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Δίδεται ενδεχομένω περισσότερη έμφαση σε θέματα που δεν ανήκουν ε, στην πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου αυτά αυτά. Και έτσι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ε, δούριος ύπος. Πολλής λόγος γίνεται για την παρουσίαση της εργαλειοθήκης, τα μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου. Τώρα, όλοι βέβαια γνωρίζουμε ότι ορισμένοι αγρότες επιλέγουν πολύ επικίνδυνες στρατηγικές αξιοποιώντας τις ευκαιρίες ε, της αγοράς που μπορεί να τους ωφελήσουν ιδιαίτερως μία στιγμή σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε ανάληψη υπερβολικού κόστους ή υπερβολικού κινδύνου σε μεταγενέστερο στάδιο. Επομένως η διαχείριση κινδύνου λειτουργεί ως ασφαλιστική ε, δικλίδα. Ότι δηλαδή ε, στην, όταν... Ε, δηλαδή, όταν είναι οι συνθήκες ευνοϊκές, μπορεί ο αγρότης να αναλάβει αυτό το ρίσκο, όταν είναι λιγότερο ευνοϊκές ε, θα χαίρει στήριξη. Ε, έχει θεσπιστεί αυτό, αυτή η έννοια του ηθικού κινδύνου, ο οποίος λειτουργήσε τόσο καταστρεπτικά στον τραπεζικό τομέα. Και πολλά είναι τα επιχειρήματα που μπορούν να προβληθούν εναντίον αυτής της κατάστασης. Η στήριξη του εισοδήματο που εντάσσεται στον πυλώνα 1, ε, ιστορικά πάντοτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ως στόχο να προστατεύσει τους αγρότες από, την, ε, ε, από το ευμετάβολο των αγορών παγκοσμίω. Και τώρα έχουμε πάλι πολιτική στον πυλώνα 1, ε, τις πληρωμές, αλλά αυτά πάνε στον δεύτερο πυλώνα. Νομίζω ότι η προτεραιότητα αυτή θα πρέπει να διαγραφεί, γιατί μας οδηγεί σε ολισθηρό δρόμο. Πολύ προσοχή δίνεται στην ε, μεταβίβαση της γνώσης, στην καινοτομία. Δεν λειτουργεί πολύ καλά η μεταβίβαση της γνώσης, ούτως ώστε να προκαλέσει, ε, ε, να δημιουργήσει καινοτομία καινοτομία. Οι υπερβολικές κανονιστικές ρυθμίσεις είναι αυτό το οποίο μπλοκάρει την καινοτομία και θα πρέπει σε αυτό το επίπεδο να δράσουμε. Υπάρχουν εθνικά ε, κανονιστικά ρυθμιστικά σχέδια τα οποία αυτά είναι τελικά που λειτουργούν ως τροχοπέδι για τη διάδοση και την ενίσχυση της καινοτομία. Και μια τρίτη προτεραιότητα που περιλαμβάνει η πρόταση αυτή είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αναφέρεται μάλιστα ρητός ανταγωνιστικότητας όλων των ειδών αγροτικής δραστηριότητας. Και εδώ έχουμε ένα δούριο υποπραγματικά, διότι μπορεί κανείς να προβάλλει το επιχείρημα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν προς όφελος της επάρκειας ε, τροφίμων που ενισχύουν την αηφορία, που έχουν θετικές επιπτώσεις στην εδαφική συνοχή. Αλλά έχουμε και, άλλες, ε, ε, και άλλα δραστηριότητες ε, τα οποία ουσιαστικά απειλούν την αηφορία, την εδαφική συνοχή κτλ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί ο πυλώνας υπαριθμών 2 θα πρέπει με αδιαφοροποίητο, με αδιάκριτο, αν χωρίς διακρίσεις τρόπο να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα όλων των ειδών αγροτικής δραστηριότητας, γεωργικής δραστηριότητας. Και θέλω αυτό να το στηρίξω με στοιχεία τεχνικά που έχουν προκύψει από μια έρευνα στις ε, κάτω χώρες. Έχουμε το, τη γεωργία χαμηλού κόστους από τη μία και τη γεωργία υψηλής τεχνολογίας από την άλλη. Ένας άνθρωπος κάνει όλη τη δουλειά και θα πρέπει οι δύο, τα δύο είδη γεωργικής δραστηριότητας να ε, οδηγούν ακριβώς το ίδιο εισόδημα. Στην αγροτική εκμετάλλευση υψηλής τεχνολογίας χρειαζόταν για παράδειγμα 800.000 ε, τόνοι γάλακτος το χρόνο για να ε, δημιουργηθεί το ίδιο εισόδημα. Ενώ ε, στην ε, τεχνολογία χαμηλού κόστους το 50%. Τα μισά λίτρα γάλακτος χρειάζονταν για να δημιουργηθεί το ίδιο εισόδημα. Αφού το αγρόκτημα υψηλής τεχνολογίας είχε ε, τα διπλάσια ε, κόστη, γιατί ήταν διπλάσιο σε μέγεθος από το αγρόκτημα χαμηλού κόστους, γι' αυτό τελικά το εισόδημα ήταν το ίδιο. Μιλούμε για 36 ευρώ για ανακυλό γάλακτος και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα ε, τελείως διαφορετικό καθεστώς τιμών. Οι τιμές έχουν κατρακυλήσει και υπάρχει πολύ μεγάλη διακύμανση οι τιμές κατέβηκαν στα 24 από τα 36 και σε αυτή την περίπτωση ε, το αγρόκτημα υψηλής τεχνολογίας ξαφνικά έχει αρνητικές ταμιακές ροές και ε, αμέσως αντιμετωπίζει μια οξία κρίση ενώ το αγρόκτημα χαμηλού κόστου συνεχίζει να παράγει. Στην περίπτωση δηλαδή ε, της κατρακύλας των τιμών παραγωγού. Ε, αυτά τα είδαμε και στα αγροκτήματα στα οποία ερευνήσαμε, αλλά το έχουμε δει και στην πράξη. Δεν θέλω να μπω σε όλα αυτά τα τεχνικά στοιχεία και σε λεπτομέρειες. Όμως τα δεδομένα που έχουμε, εμπειρικά δεδομένα, έχουν δείξει ότι πριν από την τρέχουσα κρίση οι μικρές ε, αγροτικές εκμεταλλεύσεις κερδίζουν περισσότερο αναλύτρο γάλακτος και άρα έχουν υψηλότερες αποταμιεύσεις από τις ε, υψηλής εντάσεως ε, αγροτικές εκμεταλλεύσεις. από 8 στα 3 ευρώ ανά εκατοστό λίτρο γάλακτος. Επομένως, τα θετικά ε, στοιχεία σε μια προηγούμενη κατάσταση μη κρίσης είναι αυτά που δημιουργούν και την περισσότερη ευαισθησία σε περίπτωση κρίσης. Μη διαφοροποιημένες προτεραιότητες, Ουσιαστικά οι αγροτικέ εκμεταλλεύσεις υψηλή τεχνολογίας διατρέχουν τον κίνδυνο να στοιχηματίσουν στο λάθος, στο κουτσό άλογο αν θέλετε. Βεβαίως υπήρξαν ε, αντιδράσεις, προσπάθειες ε, απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή προσπάθεια παραγωγής προϊόντων με περισσότερη προστιθέμενη αξία, διαφοροποίηση, το αγρόκτημα λειτουργεί και ως πηγή παραγωγής ενέργειας, ε, το αγρόκτημα προσφέρει νέες υπηρεσίες, βασίζεται σε μία νέα σειρά πόρων. Δηλαδή, μιλούμε για τις πολυλειτουργικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Είναι ένα πρότυπο το οποίο διαδίδεται παντού στην Ευρώπη και αναγνωρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα που ψήφισε το 2010. Το σημαντικό όμως είναι το εξή. Ορισμένοι στην αρχή θεωρούσαν ότι οι πολυλειτουργικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα λειτουργήσουν αρνητικά ως προς την παραγωγή τροφίμων. Και έχουν γίνει πολύ σημαντικές έρευνες στην Ιταλία, οι οποίες δείχνουν ότι τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, πολυλειτουργικοί αγρότες, αν θέλετε, επένδυσαν πολύ περισσότερα, ε, έχουν κάνει πολύ περισσότερες επενδύσεις στην παραγωγή τροφίμων συγκριτικά με αυτούς που καλλιεργούσαν ένα μόνο πράγμα ή που εξέτρεφαν ένα μόνο ε, είδος ε, στην κτηνοτροφική του δραστηριότητα. Στις κάτω χώρες ε, έχουμε ακριβώς τα ίδια στοιχεία, ε, τα ίδια πορίσματα. Η πολυλειτουργική γεωργική δραστηριότητα στηρίζει την παραγωγή τροφίμων και δεν την απειλεί καθόλου. Και όλα αυτά δείχνουν ότι είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί ακόμα περισσότερο αυτό το εγχείρημα των πολυλειτουργικών ε, αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέσω της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Είναι σημαντικό αυτό όχι μόνο για την γεωργία αυτή καθεαυτή, αλλά διότι η πολυλειτουργικότητα επηρεάζει πολύ θετικά την ύπεθρο γενικότερα. Η αντίληψη που έχουν οι κάτοικοι για την ποιότητα της ζωής τους. Αυτή εξαρτάται και διαμορφώνεται από την αντίληψη που έχουν για το κοινωνικό κεφάλαιο στην ίδια περιοχή. Και αυτή η ε, ποιότητα εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη μη πολυλειτουργικών ε, γεωργικών δραστηριοτήτων. Η πολυλειτουργική γεωργία προσφέρει υπηρεσίες, προσφέρει σημεία συνάντησης, δημιουργεί νέες αγορές όπου συναντώνται ε, οι αγρότες τοπικά με τον υπόλοιπο τοπικό πληθυσμό. Επομένως και σε επίπεδο αγροκτήματος αλλά και σε, όλη την ύπεθρο γενικότερα αυτού του είδους η δραστηριότητα, η πολυλειτουργική είναι εξαιρετικά σημαντική και θα πρέπει να στηριχθεί ακόμα περισσότερο. Και όπως είπα και προηγουμένως, για να επιτευχθούν όλα αυτά ε, ε, έχουν συσταθεί ομάδες παραγωγών, έτσι όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 της πρότασης. Οι ομάδες παραγωγών είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Βλέπετε τρεις νέους αγρότες από ε, το βόρειο μέρος στις κάτω χώρες. Ήταν μέλη ενός εδαφικού συνεταιρισμού, ο οποίος ήταν πολύ δραστήριο στην διατήρηση του τοπίου εκεί και σε συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα. Δεν είναι εξαίρεση αυτό και στη Γερμανία έχουμε αντίστοιχες ομάδες παραγωγών και στην Ιταλία ε, και έχουμε και αντίστοιχες ζώνες και περιοχές όπου γίνεται προσπάθεια ε, παρόμοιες λειτουργίας και στην Πορτογαλία το ίδιο έχουμε τοπικές οργανώσεις για τη διαχείριση ε, του εδάφους της επικράτειας σε τοπικό επίπεδο. Αυτή η συγκεκριμένη ομάδα, αλλά και πολλές άλλες, έχει βελτιώσει ιδιαιτέρως την αηφορία της δραστηριότητάς της. Μέσα σε λίγα χρόνια κατάφεραν να ε, περιορίσουν δραστικά το επίπεδο των εκπομπών τους, για παράδειγμα, και των εκκλήσεων. Είναι ε, πολύ ενεργοί προσπαθώντας η γεωργική δραστηριότητα να εξαρτάται όλο και λιγότερο από εξωτερική συμβολή Δηλαδή, μιλούμε για μια γεωργία χαμηλού κόστους και χαμηλής εισαγωγής, αν θέλετε, ένας κύκλος που είναι αυτοθοτροφοδοτούμενος και έτσι καλύπτονται περισσότερο οι ανάγκες του ε, πληθυσμού. Αυτές οι ομάδες παραγωγών ε, είναι εξαιρετικά σημαντικές. Θα πρέπει σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης να μην προβλέπονται εντελώς καινούρια ρυθμιστικά σχέδια και προγράμματα, αλλά θα πρέπει η διοίκηση σε τοπικό ή κεντρικό επίπεδο να προσπαθήσει να κάνει τη σύνδεση με, την, τα ήδη υφιστάμενα εργαλεία, θεσμικά εργαλεία. Τώρα, ε, ποια σημεία επιδέχονται βελτίωσης ε, στην πρόταση αυτή. Σε όλη την Ευρώπη απευθύνεται αυτή η έκκληση για ελάφρυνση του διοικητικού άχθους, όπως ε, και με τον πυλώνα όπου όσοι έχουν λαμβάνει λιγότερο, λιγότερα από 5.000 ευρώ ε, δεν χρειάζεται να ε, ε, συμμορφούνται με πολύ επαχθείς διοικητικές προϋποθέσεις. Και στον πυλώνα 2 θα μπορούσε να προβλεφθεί αυτό με τα 50.000 ευρώ ή με τα 5 ή 10.000 ευρώ για να μπορέσουν περισσότεροι να δρέψουν τα ωφέλη της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Να μειωθεί δηλαδή το διοικητικό άχθος, ο διοικητικός φόρτος. Από εκεί και πέρα η αξιολόγηση χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων. Να περιλαμβάνει η αξιολόγηση και τις διαδικασίες, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί εύρυθμα, ε, εφαρμόζεται εύρυθμα η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και η πιο σημαντική σύσταση, αυτό το οποίο χρήζει περαιτέρω βελτίωσης, είναι η σύνδεση, η άρρηκτη σύνδεση μεταξύ των κοινών δραστηριοτήτων από την μία και των επενδύσεων πάνω στο αγρόκτημα αυτό καθεαυτό από την άλλη. Έχουμε το άρθρο 18 το άρθρο 20 ε, για την ανάπτυξη την επιχειρηματική των αγροκτημάτων. Μετά έχουμε τις κοινέ δράσεις ε, που άρθρο 17, βασικές υπηρεσίες το άρθρο 21, ομάδες παραγωγών στο άρθρο 28. Όλα αυτά, ε, κάθε άρθρο αναφέρεται σε ξεχωριστό στοιχείο, αλλά θα πρέπει να συνδέονται όλα αυτά και μάλιστα με έξυπνο τρόπο. Γιατί, Γιατί αυτή τη στιγμή πώς έχει κατάσταση σε πολλά σημεία στην Ευρώπη. Οι αγρότες μπορεί να συνδυάζουν την αγροτική δραστηριότητα μαζί με την πώληση και μπαίνουν σε ένωση ή σε συνεταιρισμό και ξεκινούν να πουλούν τα δικά τους προϊόντα αλλά και των άλλων, ο ένας του άλλου δηλαδή τα προϊόντα. Αυτό είναι καλό για τον καταναλωτή γιατί διευρύνεται η γάμα προϊόντων που προσφέρεται σε συγκεκριμένη αγροτική εκμετάλλευση και για τον αγρότη είναι αυτό πολύ σημαντικό γιατί μπορεί πλέον να πουλήσει πολύ περισσότερα. Ε, αξιοποιείται το διαδίκτυο ε, οι αυτοματοποιημένοι τρόποι επίτευξης ισορροπίας. Επίσης, ο αγρότης υπ' αυτή την έννοια μπορεί να φτάσει σε πολύ πιο απομακρυσμένες περιοχές. Έχουμε δηλαδή μια κυκλική διάρθρωση η οποία αναπτύσσεται και εμφανίζεται σε πολλά σημεία στην Ευρώπη και βρίσκεται σε αντίθεση με την ε, κλασική διάρθρωση του σούπερ μάρκετ το οποίο δεν λειτουργεί ε, ακτινοτά. Εδώ λοιπόν μπορούμε να έχουμε προϊόντα που έρχονται από το βορρά, ε, φτάνουν σε ένα κέντρο, διανομή στο κέντρο ε, και μετά ξαναπηγαίνουν στο βορρά. Το σούπερ μάρκετ λοιπόν ε, μπορεί να λειτουργήσει ακτινοτά και όχι κυκλικά και έτσι έχουμε περισσότερο πηγενέλα προϊόντων μπορούν να αποφευχτούν αυτά και να επιλεγεί ο κύκλος, η κυκλική διάταξη. Για να επιτευχθούν όλα αυτά χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας, για την κοινή θέση σε εμπορία, τις κοινέ δράσεις marketing, για την καλύτερη προσβασιμότητα, για τη δημιουργία δομών ε, στήριξης και υποδομής Μπορούν λοιπόν οι επενδύσεις στο αγρόκτημα να συνδυαστούν με τις κοινέ δράσεις. Και ε, θα πρέπει να υπάρχει μια διάταξη σε κάποιο άρθρο της πρότασης που να το καθιστά αυτό σαφές. Να ζητά υψηλότερα επίπεδα στήριξης όταν δημιουργούνται αυτές οι συνέργειες και αυτοί οι συνδυασμοί. Έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση μεταξύ καταναλωτών από τη μία και παραγωγών από την άλλη. Έχουμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 8 Ιουλίου του 2011 και εκεί γίνεται λόγος για ε, τοπικά ε, εργαλεία, ε, τοπικά δυναμικά εργαλεία. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και μάλιστα στην πράξη. Αυτά είχα να πω μέχρι αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, Ζων. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση, η διαχείριση του κινδύνου στο δεύτερο πυλώνα, καθώς και οι άλλες παρατηρήσεις σου, που εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας πολύ μας ενδιαφέρουν τα πράγματα αυτά. Λοιπόν, τώρα θέλω να γίνει μια συζήτηση. Αρχίζουμε από την κυρία Κέστιγκερ και ε, εν συνεχεία θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντόρφαν. Ελίζαμπεθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εξηγήσεις. Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον δύο οι προκλήσεις που ίσως δεν ε, συζητούνται επαρκώς. Αυξάνουν οι τιμές διότι αυξάνει και η ζήτηση στις αναπτυσσόμενες χώρες για λύπη και για άλλες ουσίες. Το ίδιο οι εξαγωγές δεν είναι πάντα βέβαιον το ύψος τους λόγω διαφόρων κυκλικών διαφορών. Και στο κείμενο δεν βρίσκουμε όμως ε, απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Κάτι άλλο το οποίο μου φαίνεται ότι δεν εξηγείται παρκώς είναι των φορέων, των ορυκτών φορέων ενέργειας και τη εξάρτηση στην οποία τελούμε εδώ στην Ευρώπη από τους φορεί αυτούς. Ενώ έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και ολική ενέργεια και ε, την ε, βιομάζα που θα ωφελήσουν και τις αγροτικές μας εκμεταλλεύσεις. Υπάρχουν λοιπόν εδώ ορισμένοι τομείς που είναι ελπιδοφόροι και που πρέπει να διευκρινιστούν και το screening στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμο και νομίζω ότι και η Επιτροπή Γεωργίας έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα αυτό, δηλαδή η έλεγχη μπορεί να είναι και προβληματική. Δηλαδή σε πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν ήδη κάνει σημαντικά πράγματα οι γεωργοί για το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτοί οι γεωργοί θα δουν να επιδεινώνεται η κατάστασή τους μετά από τις νέες προτάσεις της Κομισιόν. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Με ενδιαφέρει επίσης Αυτός ο καθορισμός των 25% των κονδυλίων για προγράμματα που περιλαμβάνονται μόνο στο αιτιολογικό. Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα έχει και περαιτέρω επιπτώσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιδίνω της θέσης τους στις χώρες μέλη. Για τις έξι προτεραιότητες τώρα, νομίζω τα εξηγήσατε πράγματι και εν εκτάση. Για το πρώτο, για τη μεταφορά γνώσης και καινοτομία στην Γεωργία, εδώ πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση όταν μιλούμε για την κατανομή των κονδυλίων. Η μεταρρύθμιση αυτή απευθύνεται κυρίως στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αλλά η παραγωγή τροφίμων δηλαδή δεν είναι ο κεντρικός παραλήπτης. Εδώ χωρούν και διαφορετικές ερμηνείες και γι' αυτό χρειάζεται μια διευκρίνηση. Ποιος καθορίζει την έννοια, οι χώρες μέλη ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η βελτίωση τώρα της ανταγωνιστικότητας όλων των ειδών γεωργίας. Και εδώ μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό να λεχθεί εάν καλύπτονται όλοι οι τομείς ή εάν θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος για ορισμένους τομείς που χρειάζονται επιγόντως ενίσχυση. Μιλήσατε και για την σημασία των οργανώσεων παραγωγών και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι συνεταιρισμοί και μάλιστα θα έπρεπε να είχε αρχίσει και πολύ νωρίτερα. Για το θέμα των δικημάνσεων τιμών που είπατε κι εσείς, ελάχιστα θίγεται μόνο την ασφάλιση έναντι των κινδύνων, που για ορισμένε χώρε μέλη δεν θα είναι και το σωστό εργαλείο για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Πιστεύω ιδίω ότι ο δασοκομικό τομέα δεν λαμβάνεται παρκώ υπόψη στι προτάσει, στα υποβληθέντα κείμενα δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι και οικονομικά εδώ κρύβεται τεράστιο δυναμικό για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για τις ανανεώσιμες ενέργειες, δηλαδή όπως είπαμε και στην αρχή, και που ακόμα μένουν πολλά να γίνουν. Με ενδιαφέρει ακόμη ένα θέμα. Οι νέοι αγρότες που έχουν ιδιαίτερη θέση σε αυτή την ανανέωση και με την πρόταση μέτρων στον πρώτο πυλώνα που υποτίθεται ότι θα ωφελήσουν ιδιαίτερα και θα ευνοήσουν τους ε, νέους αγρότες που σε ένα μεγάλο ποσοστό αναλαμβάνουν δραστηριότητα για πρώτη φορά. Ποιες άλλες προτάσεις μπορούν να γίνουν και μέτρα να ληφθούν για να υπάρχουν και στο μέλλον αυτοί που θα ηγηθούν των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ευχαριστώ, Ελίζαμπετ. Χέρμπερτ. Και μετά ο Αντιπρόεδρος. Ντόρφμαν. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Πρώτη, κύριε καθηγητά, είπατε σωστά τι θα γίνει με το risk management. Δεν νομίζετε κι εσείς ότι το εργαλείο αυτό έχει καταλήξει εν τέλει σε λάθος πυλώνα, δηλαδή αυτή η διαχείριση κινδύνου που έχει σχέση ε, βέβαια με τις τιμές και το εισόδημα των αγροτών, κατά τη γνώμη μου, είναι καθαρά, είναι κλασικό ε, στοιχείο του εισοδήματο και θα έπρεπε να μπει στον πρώτο πυλώνα, όπως και προβλέπει το άθρο 68. Δεν νομίζετε επίσης ότι αυτό πρέπει να το σκεφτείτε, αν ίσως αυτό το εργαλείο Διαχείριση του κινδύνου θα έπρεπε να τοποθετηθεί αλλού. Για το greening, το πρασίνισμα, δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συμφωνώ με τα όσα είπε και η κυρία Κρέστιγκερ. Είπατε ότι το πρασίνισμα είναι λογικό και για τους δύο πυλώνες. Εγώ θα προσθέσω, δεν ξέρω αν είναι λογικό, αν ήταν λογικό θα έπρεπε να, είναι, να μην είναι τουλάχιστον απόλυτα ανεξάρτητο όπως ήταν μέχρι τώρα στις προτάσεις θα έπρεπε να προβλέπετε τουλάχιστον ότι κάθε εκμετάλλευση του δεύτερου πυλώνα να κάνει να λαμβάνει μέτρα για το πρασίνισμα μέσω των περιβαλλοντικών προγραμμάτων ώστε αυτό το πρασίνισμα του δεύτερου πυλώνα να είναι η προϋπόθεση και το πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα. Γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να έχουμε επικάλυψη και επικάλυψη και ελέγχων δεν νομίζετε ότι μπορούν να διασυνδεθούν καλύτερα, θα έπρεπε μάλλον να διασυνδεθούν καλύτερα τα πράγματα μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόλσεν και μετά ο Μάρτιν Όσλι. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο πρόγραμμα LEADER. Πρέπει να υποφεληθούμε από όλες τις δυνατότητες ε, των ε, γεωργικών ζωνών. Θα πρέπει να υποστηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες και παράλληλα να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ διαφόρων κρατών μελών και διαφορετικών περιοχών και περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια λεπτομέρεια, αλλά σημαντική, κατά γνώμη μου. Μετά από αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να αναφερθώ και στην ευημερία των ζώων. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τις προκλήσεις. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί, η γεωργία. Οι γεωργοί πρέπει να παράγουν α, τρόφιμα. Προωθούν τη βιοπικιλότητα. Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ευημερία των ζώων. Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κλίμα. Ο Γιώργος θα πρέπει να παράγει ίσως τη δική του ενέργεια. Να διάφορες λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ούτως ώστε η γεωργία να είναι αποδοτική. Και οικονομικά και κοινωνικά. Νομίζω ότι η δημιουργία δικτύων διανομής με συνεταιρισμούς, με οργανώσεις, ό,τι όνομα και να θέλετε να δώσετε αυτές τις οργανώσεις. Αυτό πρέπει να γίνει. Είναι σημαντικό. Ε, προέρχομαι από μια χώρα που υπάρχουν πολύ μικροί ε, επιχειρηματίες ε, που πάνε μια χαρά. Που φτιάχνουν τυρί, δέχονται τουρίστες και παράλληλα ασχολούνται με τη διανομή και την πώληση αυτού του τυριού. Για όλη αυτή τη δουλειά δεν αρκούν 24 ώρες της μέρας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιες εταιρισμοί, τέτοιες οργανώσεις, τέτοιοι όμιλοι αν θέλετε γεωργών. Και επανέρχομαι σε κάτι που μου αρέσει να λέω συχνά τις δυνατότητες χρηματοδότησης νέων ιδεών στις ε, περιοχές της υπαίθρου. Υπάρχει σήμερα οικονομική κρίση, η χρηματοπιστωτική κρίση που αφορά όλους πια. Υπάρχει και η τραπεζική κρίση που ε, απειλεί την ανάπτυξη της υπαίθρου. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να δανειστεί κανείς από τις τράπεζες. Λοιπόν, χρειάζομαστε ε, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που θα μας επέτρεπαν σε κάποιο βαθμό να σταθεροποιήσουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης της περιοχής της Υπέθρου. Ευχαριστώ. Μάρτιν. Και μετά Γκαρσία Περέθ. Λίγα σύντομα σχόλια. Συμφωνώ την άποψή σας υπέρ της πολυλειτουργικής γεωργίας και ίσως και μάλλον με την έρευνά σας καταστήσατε σαφές ότι μια γεωργία που βασίζεται σε περισσότερα θεμέλια, σε πλείονα θεμέλια, σε περισσότερα πόδια, είναι βέβαια πιο ανθεκτική και στις κρίσεις. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να το προβάλλουμε, ιδιαίτερα και στη δημιουργία του δεύτερου πυλώνα. Όχι μονάχα χρήματα του δεύτερου πυλώνα σε ένα πυλώνα επενδύσεων που θα οδηγήσουν σε μια τεχνικοποίηση της ε, ε, γεωργίας, αλλά σε μια πολυλειτουργική γεωργία. Αυτό που βρήκα ενδιαφέρον και συμφωνώ με τη γνώμη σας είναι που είπατε ότι η εξασφάλιση κατά των κινδύνων στο δεύτερο πυλώνα δεν μπορεί να αποτελέσει εργαλείο το οποίο θα πρέπει να επιδιώξουμε. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί σωστά είπατε ότι δεν μπορεί κανείς να ιδιωτικοποιεί τα κέρδη και να φορτώνει στην κοινωνία εν τέλει τις ζημίες. Θεωρώ λοιπόν και εγώ, όπως και εσείς, ότι αυτή αυτός ο τρόπος διασφάλισης στον δεύτερο πυλώνα δεν έχει απολύτως καμία θέση. Εάν θέλουμε εξασφάλιση έναν των κινδύνων πρέπει να σκεφτούμε κάποια άλλα μοντέλα. Αλλά ε, να μην παραφορτώσουμε το δεύτερο πυλώνα. Κάτι που μου φάνηκε να λείπει είναι για τα, με, τα αγροτικά μέτρα περιβάλλοντος, ας το πω έτσι. Εκεί πρέπει αυτά να ενταθούν στον δεύτερο πυλώνα και να θέσουμε και κριτικά ερωτήματα διότι τα μέτρα δεν έχουν ακόμη επιτύχει τα αποθητά αποτελέσματα. Άλλωστε και το ελεγκτικό συνέδριο ρωτά εάν κάποια μέτρα είναι όντως σκόπιμα, εάν ίσως είναι απαραίτητη κάποια διαφοροποίηση των μέτρων και μάλλον ένας προσανατολισμός προς μια οικολογική γεωργία που θα ήταν περισσότερο Νομίζω ότι κάποια τέτοια μέτρα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο. Κάτι που με εκπλήσει και που το δείξατε στην πρώτη σας διαφάνεια είναι που είπατε ότι η άρση της δομής των αξώνων είναι καλή. Πώς το αιτιολογείτε αυτό. Νομίζω ότι η δομή αυτή με τους άξονες σε, πολλούς χώρες, έχει, σε πολλές συγγνώμη, χώρες έχει αποδείξει την αξία της και έχει διασφαλίσει ότι τα χρήματα θα δίνονται σε διάφορες χώρες μέλη προς κάθε κατεύθυνση. Εάν εγκαταληφθεί αυτή η δομή των αξώνων θα υπάρχουν ορισμένες χώρες μέλη οι οποίες θα κατευθύνουν μέτρα προς ορισμένους, ορισμένους μονοτομείς και για παράδειγμα τα αγροτικά περιβαλλοντικά μέτρα δεν θα τα ενισχύουν. Γιατί δηλαδή χαιρετίζεται το γεγονός ότι καταλείπονται οι άξονες. Ναι μεν 25% ακόμα δεν έχουν ε, οριστικά κατανεμηθεί αλλά αυτά τα 25% για τα αγροτικά περιβαλλοντικά μέτρα θα πρέπει να είναι το απόλυτο ελάχιστο. Κατά τη δική μας δε γνώμη θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερα. Για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας θα πρέπει να δούμε ότι η βιολογική γεωργία είναι ένα τομέα που υπόσχεται πολλά και υπάρχει και μια αγορά για τα προϊόντα αυτά. Θα ήταν κατά βάση λάθος για την περαιτέρω εξέλιξη, να μην χρηματοδοτεί περισσότερο ο τομέας αυτός. Και, κάτι, και ένα τελευταίο που νομίζω πρέπει να δοθούν περισσότερα, ε, να δοθούν περισσότερα κονδύλια είναι τα προγράμματα leader. Εγώ θεωρώ ότι αυτά πρέπει να προβληθούν και να εμφανιστούν στο προσκήνιο ακόμα εντονότερα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και να μην επαναλάβω τα ερωτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοι, με τα οποία συμφωνώ απολύτως βέβαια. Μία από τις προκλήσεις που υψώνονται μπροστά μας στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή αγροτικής πολιτικής είναι η βιωσιμότητα, η φορεία της υπαίθρου. Όλοι γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση διαβιούν διάφορες ε, περιοχές αγροτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διατρέχουν το κίνδυνο ε, πλήρους εξαφάνισης αν θέλετε εάν δεν λειτουργήσει αυτή η μεταρρύθμιση και δεν καταφέρει να κρατήσει τον κόσμο στην υπαίθρο. Εξού λοιπόν και οι τοποθετήσει ε, που παρουσιάστηκαν από τον ε, κύριο καθηγητή. Ήταν πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι παρατηρήσεις. Η καινοτομία, η αντιγωνιστικότητα, το περιβάλλον θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της μεταρρύθμισης της πολιτικής της υπαίθρου. Βασικό θέμα στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα είναι να εγγυηθούμε το εισόδημα των αγροτών. Από την άλλη όμως, αν δεν καταφέρουμε να δουλέψουμε και το άλλο επίπεδο του συνδυασμού και του συντονισμού δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Επομένως, δύο είναι αυτά που μας ανησυχούν κατά βάση ως προς τη μεταρρύθμιση και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Πρώτον, η σχέση με τους νέους. Και έγινε αναφορά σε αυτό. Δυστυχώς, δεν έχουμε καταφέρει να προσφέρουμε κίνητρο και να στηρίξουμε τους νέους που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του αγρότη, που νιώθουν οι ίδιοι την επιθυμία και νιώθουν, ε, ε, την, έχουν το κίνητρο να ασχοληθούν με αυτά. Δεν τους έχουμε στηρίξει επαρκώς. Από εκεί και πέρα ε, εξαφάνιση της βοήθειας λόγω της διακοπής της δραστηριότητας λόγω του ότι θα διακοπεί η ενίσχυση αυτή στο μέλλον. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή οι νέοι ε, που έχουν την ε, επισημία να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα δεν ε, μπορούν να τύχουν επαρκού στήριξη. Θα πρέπει να το αντισταθμίσουμε αυτό με άλλα μέτρα. Και Ω προ την ανταγωνιστικότητα, καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη μας την διαφοροποίηση στη γεωργική δραστηριότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ίσως εξαφανιστούν οι ενισχύσει ε, σε επενδύσεις σε αρδευτικά έργα βάσει του κλίματος που επικρατεί σε ορισμένες χώρες ή περιφέρειες. Το κλίμα και η ύπαρξη αρδευτικών καναλιών είναι αυτά από τα οποία εξαρτάται απολύτω η γεωργική δραστηριότητα και η εκτινοτροφία δραστηριότητα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διατηρηθούν αυτά τα εργαλεία, επενδύσει σε αρδευτικά έργα, ε, γιατί αλλιώ θα εξαφανιστεί η ακροτική δραστηριότητα στι περιοχέ που εξαρτώνται από την ε, ε, ύπαρξη άρδευση. Από εκεί και πέρα και πολλέ άλλε ερωτήσει έχω να θέσω, αλλά τι έχουν ήδη θέσει οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Νικουλέσκου και μετά ο Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσίαση που ακούσαμε. Υπάρχουν τρία πράγματα που με ανησυχούν και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, θα συμφωνήσουμε από αυτόν. Καταρχάς, δεν μπορούμε να έχουμε γεωργία χωρίς ε, αγρότες, χωρίς γεωργούς. Ε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεύτερον, μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα της α, ε, γεωργικής δραστηριότητας και τις καλά ε, διασυνδεδεμένες αγορές. Υπάρχουν ε, αγορέ ε, οι οποίε είναι απομονωμένε όχι γιατί είναι μεγάλε οι αποστάσει από το κέντρο, ας πούμε, αλλά γιατί υπάρχουν προβλήματα υποδομών. Επίση θα πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση των προτεραιοτήτων. Δεν υπάρχουν αρκετέ επενδύσει στι υποδομέ. Και δεν μπορούμε να έχουμε μοντέρνε εκμεταλλεύσει αν δεν έχουμε μοντέρνες υποδομέ. Και αυτό είναι το πρόβλημα σε πολλέ από τι νέε χώρε μέλη. Στον άλλο σημαντικό πυλώνα, τον πρώτο πυλώνα, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι νέοι ε, γεωργοί εγκαθίσταται στην ε, Ήπεθρο, αλλά για να εγκατασταθούν θα πρέπει να έχουν ένα μοντέρνο περιβάλλον που να τους πλαισιώνει. Να ζουν μέσα σε ένα μοντέρνο περιβάλλον, δηλαδή νερό μέσα, που δεν περνάει μέσα από ε, τους σωλήνες, ε, να μην είναι απλώς τραχούμενο, ε, ίντερνετ υψηλής ποιο, ε, ταχύτητας κτλ. Λείπουν τέτοια πράγματα από τις περιοχές υπαίθρου και θα πρέπει να τα εξασφαλίσουμε. Ο αντιπρόεδρος Ακεριέση και μετά ο Τζιμ Νίκολσον. Ευχαριστώ. Η ανάπτυξη υπαίθρου. Πώς ορίζεται την ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα ήθελα να το μάθω αυτό, θα ήθελα να το καταλάβω. Είναι η ανάπτυξη της γεωργίας. Είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου. Είναι η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία. Είναι το περιβάλλον. Τι είναι από όλα αυτά, τι ισχύει από όλα αυτά. Εγώ νόμιζα ότι η ανάπτυξη υπαίθρου ήταν κάτι άλλο. Είναι η προσαρμογή σε κάποιες προσδοκίες. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό... Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες του 40% του πληθυσμού. Οι υπουργοί προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το δεύτερο πυλόν από ό,τι ξέρω για επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της γεωργίας. Και υπάρχει μια μόδα υπέρ του πρασινίσματος από ό,τι βλέπω και της καινοτομίας. Όλοι έχουν κολλήσει σε αυτή τη λέξη καινοτομία και την πιπιλίζουν. Γιατί κάπου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί δηλαδή για να πληρώνει την περιβαλλοντική προστασία. Αυτά είναι λεφτά που πρέπει να πάνε στους γεωργούς. Το πρασίνισμα αποδυναμώνει την ανταγωνιστική γεωργία. Ε, δεν την κάνει λιγότερο ανταγωνιστική. Χάνουν οι γεωργοί λόγω του πρασινίσματος. Επίσης οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Και πρέπει να το πούμε. Επίσης, πώς ξοδεύουμε για την ανάπτυξη της υπαίθρου και σε κάθε χώρα δηλαδή. Σε ποιες χώρες ξοδεύουμε τα χρήματα αυτά. Ε, για να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα, ε, γιατί έχουμε διάφορες απορίες. Και έπειτα, η σχέση ανάμεσα στην πολιτική συνοχή και το δεύτερο πυλώνα. Ανάπτυξη τη υπαίθρου δηλαδή. Ας είμαστε ειλικρινεί. Η ανάπτυξη της υπαίθρου, που είναι κάτι που θέλουμε ως Γεωργή, είναι στην πολιτική συνοχή. Ε, η πολιτική συνοχή όμω εστιάζεται στη χρηματοδότηση των πόλεων, για την ανάπτυξη των πόλεων. Πού είναι η χρηματοδότηση υπαίθρου, αν η πολιτική συνοχή είναι να προωθήσει την εδαφική συνοχή, θα έπρεπε χρηματοδοτικά πώς να αντανακλά και την ε, επιφάνεια που καλύπτει η ύπεθρος. Θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι η γεωργία, τι είναι η ανάπτυξη πέθρου, τι είναι περιβάλλον. Όλα αυτά είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα στο καλάθι της ΚΑΠ και να πούμε οι γεωργοί παίρνουν όλα αυτά τα λεφτά και παρόλα αυτά είναι άπλιστοι και θέλουν παραπάνω. Δεν είναι περίεργο που δεν τα πάνε καλά οι γεωργοί. Πώς θα μπορέσουν να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι του ανταγωνισμού όταν του αντιμετωπίσουμε έτσι. Ευχαριστώ τον κύριο Σεκυριέσκη. Jim Colston. Ευχαριστώ. Εγώ όπως ξέρετε προέρχομαι από το Ενωμένο Βασίλειο. Έχω λοιπόν κάποια ανησυχία σχετικά με το, το μέλλον, ποιο θα, με το ποιο θα είναι το μέλλον. Ε, τι χρήμα, τι κονδύλια θα υπάρχουν δηλαδή. Παρ' όλα αυτά έχω ορισμένε ερωτήσεις. Εγώ δεν πιστεύω και πολύ στο πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα. Έχει γίνει καμιά αξιολόγηση σχετικά με το πρασίνισμα και του πρώτου αλλά και του δεύτερου πυλώνα και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στον δεύτερο πυλώνα όπου εγώ νομίζω ότι εκεί πρέπει να εντοπίζεται το πρασίνισμα και επίσης έχει γίνει έρευνα σχετικά με την απλούστευση της γραφειοκρατίας η νέα πρόταση μήπως θα οδηγήσει σε περισσότερη γραφειοκρατία και λιγότερη πραγματική δουλειά επιτόπου εκεί όπου οι άνθρωποι χρειάζονται την πραγματική υποστήριξη. Έχετε λοιπόν ιδέα σχετικά με το διοικητικό κόστος. Θα αυξηθεί αυτό. Έχετε κάνει σχετική μελέτη. Εξάλλου υποστηρίζω την κυρία Πόλσεν που είπε κάτι σημαντικό. Εγώ γνωρίζω πολλούς στην περιοχή μου που δεν μπορούν να κάνουν αυτά που θα μπορούσαν να κάνουν διότι δεν λαμβάνουν έστω και μικρά δάνεια από τις τράπεζες τώρα. Και μέχρι ότου αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και φτάσουμε σε μια κατάσταση που να μπορεί να τους παρέχεται η απαραίτητη χρηματοδότηση για να αναλάβουν κάποιες από τις δράσεις αυτές. Ίσως βέβαια αυτό να γίνει, ίσως κάποια στιγμή να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση και μάλιστα δραματικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα 2-3 χρόνια. Ποιος ξέρει. Ελπίζουμε όλοι βέβαια ότι θα γίνει, αλλά επί του παρόντος και κατά πάσα πιθανότητα και στο άμεσο μέλλον βρίσκω εκεί να ε, υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία και εγώ γι' αυτό υποστηρίζω και την άποψη κυρίας Πόλσεν. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε, κύριο κύριος Άκουσα με ενδιαφέρον αυτές, είδα, είδα με ενδιαφέρον τους πίνακες με τις μικρές γαλακτοκομικές ε, ε, εκμεταλλεύσεις που βασίζονται στο βοσκοτόπι, στο γρασίδι δηλαδή και εκτρέφουν ε, μικρούς αριθμούς αγελάδων για παραγωγή γάλακτος. Και αυτό που έδειχναν οι πίνακες αυτοί, ξεκάθαρα, είναι ότι δεν μπορεί κανείς να ε, ότι το, το γάλα προέρχεται από αγελάδες οι οποίες εκτρέφονται με φυσιολογικό τρόπο. Στη Βρετανία προχωρούμε σε εντατικοποίηση της γαλακτοκομικής παραγωγής με, νέα, με παραγωγή νέων ειδών καλαμποκιού με αγελάδες οι οποίες δεν βγαίνουν στο βοσκοτόπι. Το, η ζωοτροφή τους έρχεται ε, εκεί όπου βρίσκονται μέσα και επομένως δεν έχουν και επαφή με βλαβερά ζώα. Τώρα όμως το λόμπι των πράσινων δεν χαίρεται Δεν δέχεται οι αγελάδες να είναι έγκλειστες, από την άλλη μεριά υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι αντίθετοι. εξάρω, εξάλλου η εντατικοποίηση μπορεί να γίνει μόνο στη βάση της εισαγόμενης σόγιας και ελπίζω ο Μάρτι να με ακούει. Τώρα, για τη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας. Τι είναι αυτό το τρομερό προηγούμενο με όλη αυτή τη τεχνολογία των μεταλλαγμένων οργανισμών που εδώ όμως προσφέρονται λύσεις. Αλλά τι έγινε τελικά. Ακούστηκαν τόσες ανοησίες που ενθαρρύνθηκε μάλιστα από ορισμένα κοινωτικά όργανα ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο οι άνθρωποι επενδύουν σε αυτές τις ε, νέες τεχνολογίες των ε, ε, μεταλλαγμένων οργανισμών και φτάσαμε μάλιστα και σε ένα σημείο μηδενικής ανοχής εισαγόμενης σόγιας και αυτό θα πάει ακόμα περισσότερο. Διότι στον Καναδά οι άνθρωποι είναι πολύ ευχαριστημένοι με την ε, γενετικά μεταλλαγμένη σόγια και δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τις απαγορεύσεις αυτές. Πήγα στο Ρόθαμστεντ, ερευνητικό κέντρο για γεωργικά, όπου πρόκειται να κάνουν την προσπάθεια να μεταφέρουν γνώση και να καλλιεργήσουν γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς και θα βάλουν ένα τεράστιο φράχτη, ένα τεράστιο σειρματόπλευμα γύρω από αυτό το 1,5 εκτάριο που έχουν για να μην μπαίνουν μέσα οι, ε, ε αυτοί που διαβάζουν και διαδηλώνουν. Και εσείς Μάρτιν και οι υπόλοιποι δεν είναι δυνατόν να έχετε και τα δύο. Ή θα αφήσετε τη Γεωργία να περάσει τον 21ο αιώνα στην Ευρώπη ή θα παραμείνουμε στάσιμοι μέσα σε αυτές τις απαγορεύσεις των γενετικά μεταλλαγμένων εισαγωγών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις εισαγωγικέ παρατηρήσεις στο εργαστήριο. Τέσσερις ερωτήσεις παρακαλώ. Πρώτα, η επισκόπηση αυτή με τις ε, εκμεταλλεύσεις ή υψηλής τεχνολογίας ή χαμηλού κόστους και τα σχετικά πλεονεκτήματα. συμπληρωματικά με το όσο είπε ο κ. Νικολέσκου, εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και εκμεταλλεύσεις υψηλή τεχνολογία, γιατί στο κάτω τη γραφής και οι νέοι πρέπει να επιθυμούν να συμμετάσχουν και η καλύτερη εκμετάλλευση χαμηλού κόστους είναι αυτή που μπορεί να είναι και αυτόνομη. Βέβαια αυτή οδηγείται και σε αυτοεκμετάλλευση. Ε, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα καλά τα επιχειρήματά σας στο σημείο αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Διεξάγονται εντατικέ συζητήσει, όχι εδώ στην Επιτροπή Γεωργία, αλλά με άλλου συναδέλφου μα, οι οποίοι θέλουν να περιορίσουν τα κονδύλια και για τον αγροτικό τομέα. Πώς λένε είναι δυνατόν να έχετε τα διάφορα προγράμματα δεν μπορούμε να βάλουμε όλα τα κονδύλια, να τα συνοψίσουμε όλα τα κονδύλια που δίνονται για την Ήπεθρο. Δώστε μας ορισμένα επιχειρήματα που να ενισχύσουν τη θέση μας εδώ της Επιτροπής Γεωργίας, διότι εμείς λέμε ότι είναι σημαντικό η περιοχή της Ήπεθρου να συνδιαμορφώνεται και από την αγροτική πολιτική. Τρίτο ερώτημα, ε, μετά τα όσα είπε και ο κύριος Χόισλινγκ, για τη νέα ευελιξία που περιλαμβάνεται στα νέα σχέδια, στο νέο σχέδιο κανονισμού για τη διασύνδεση των διαφόρων αξώνων που αποδυναμώνεται τώρα και επομένως θα αποφασίζουν οι περιφέρειες, οι χώρες μέλη μόνες τους με αυτόν τον τρόπο θα επενδύονται τα κοντήρια. Και τελευταία ερώτηση από τη δική σας σκοπιά. Υπάρχει μια βέλτιστη ας πούμε σχέση μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή τους και αν ναι, ποια θα ήταν αυτή η βέλτιση σχέση. Ευχαριστώ κύριε Γιάρ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον κύριο καθηγητή για τις ε, παρατηρήσεις του. Ε, λίγα σύντομα ερωτήματα. Είπατε ότι δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα εάν περιβαλλοντικά μέτρα του πρώτου πυλώνα συμπληρώνονται με περιβαλλοντικά μέτρα του δεύτερου πυλώνα. Μετά όμως είπατε, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, ότι δεν επιτρέπεται αυτό να οδηγήσει σε περισσότερη γραφειοκρατία, αλλά ότι το ζητούμενο είναι λιγότερη γραφειοκρατία. Όμως ήδη στην Κομισιόν γίνονται διαπιστώσεις ότι οι προτάσεις της Κομισιόν δεν θα οδηγήσουν σε λιγότερη, αλλά σε περισσότερη γραφειοκρατία. Επομένως κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποδεχθούμε. Εγώ είμαι βαβαρός. Στην ιδιαίτερη πατρίδα μου λοιπόν ήδη χρηματοδοτούνται πολλά περιβαλλοντικά μέτρα από, τη, από τον δεύτερο πυλώνα, για παράδειγμα η φορά. Αν όμως αυτή τώρα ενταχθεί στον πρώτο πυλώνα, πώς θα είναι δυνατόν να συνεχίσει να χρηματοδοτείται και να ενισχύεται από τον δεύτερο πυλώνα γιατί η συσφορά ε, χρηματοδοτείται στη Βαυαρία πολύ περισσότερο και προωθείται δηλαδή από τα μέτρα πρασινίσματος του πρώτου πυλώνα. Άρα θα βρεθούν σε δυσμενή θέση η Γεωργία από την άποψη αυτή. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι ναι μεν στον πρώτο πυλώνα θα πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά τα περιβαλλοντικά μέτρα του δεύτερου πυλώνα θα πρέπει να, ισχύουν επίσης και στις ε, έρευνές σας βρήκατε απαντήσεις σχετικά με το πώς θα μειωθούν οι διαφορές και οι ανισότητες στην Ευρώπη, γιατί μιλούμε για τις διαφορές στην 100 ευρώ για παράδειγμα στην Λετωνία, αλλά υπάρχουν και αλλού περιφέρειες που λαμβάνουν 600 ευρώ. Δανία για παράδειγμα, κάτω από 40 ευρώ στον δεύτερο πυλώνα. Με 40 ευρώ δεν μπορεί κανείς να χρηματοδοτήσει αγροτικά περιβαλλοντικά μέτρα, ενώ η Σλοβενία έχει 250 ευρώ στον δεύτερο πυλώνα. Ποια είναι λοιπόν η απάντηση σε αυτές τις ανισότητες, διαφορές Δεν θα ήταν σωστό να λεχθεί ότι κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να προβλέπει και να χρησιμοποιεί αλφα ποσό κονδυλίων ανεκτάριο σε κάθε, ε, στον κάθε πυλώνα. Είναι βεβαίω διαφορετικέ οι ε, καταστάσεις στις διάφορες περιφέρειες και δεν μπορούν οι Βρυξέλλες να λένε ότι όλοι οι γεωργοί θα κάνουν ακριβώ το ίδιο σε όλες τις περιφέρειες γιατί χάνεται τότε η δυνατότητα να στοχευθούν σωστά τα περιβαλλοντικά μέτρα. Το ίδιο ισχύει και για τις επενδύσεις σε ορισμένε χώρε μέλη όπως τη Γερμανία όπου ήδη έχουν γίνει σημαντικέ επενδύσει στο μέλλον δεν χρειάζονται τόσο πολλές επενδύσεις όπως στην Πολωνία για παράδειγμα ή σε νέες χώρες μέλη. Εδώ λοιπόν πρέπει να εξευρεθούν διαφορετικές απαντήσεις ώστε να αποκατασταθεί μεγαλύτερη ισότητα μέσα στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω απαντήσεις για αυτά. Επενδύουμε τώρα επίσης στο ταχύ ίντερνετ στην Ήπεθρο που είναι σημαντικό να έχουν ταχείες συνδέσεις ίντερνετ, διαδικτύου οι, ε, αγρότες. Διαπιστώνουμε στη Βαβαρία ότι σε κοινότητες όπου δεν υπάρχει ταχύ ίντερνετ δεν πηγαίνουν να εγκατασταθούν ούτε βιοτεχνίες ούτε άλλοι επαγγελματίες. Πηγαίνουν εκεί όπου έχουν πρόσβαση σε ταχύ διαδίκτυο. Χρειάζεται λοιπόν να ανοίξουμε τέτοιους δρόμους. Η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και δεν εξυπηρετείται με τον τρόπο αυτό. Πρέπει λοιπόν και αυτό να εξετάσουμε με, την, με, με τις επενδύσεις του δεύτερου πυλώνα. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι στον δεύτερο πυλώνα πρέπει να εγκατασταθούν αυτά τα μέτρα και όχι να μείνουμε μονάχα σε, μια, σε ένα είδος διαχείρισης κινδύνου. Εκεί έχει δίκιο ο Östling. το risk management κατά τη γνώμη μου πρέπει να μείνει στον πρώτο πυλώνα. Ευχαριστώ, Άλμπερ. Νταντά, μετά Κλάς και μετά θα δοθούν απαντήσεις. Ευχαριστώ. Να επανέλθω στην παρατήρηση που έκανε ο κύριος Σικιέρσκι. Γιατί το θέμα αυτό που έθεσε είναι πολιτικό, πολιτικό το ερώτημα. Η περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να ξεκινάει και να ασχολείται και να εστιάζεται μόνο στις πόλεις. Θα πρέπει ε, ως Επιτροπής ε, Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου θα πρέπει ε, να ασχοληθούμε με τις ανάγκες της Υπέθρου που δεν είναι γεωργική. Γιατί υπάρχουν σήμερα τμήματα της, Υπέθρου που δεν έχουν κανένα γεωργό. Και άλλα τμήματα της Υπέθρου που είναι εντελώς γεωργικά. Αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι ταυτόσιμα πια. Δεν θα πρέπει να τα μπερδεύουμε. Όταν κοιτάω τον κατάλογο των μέτρων που μας προτείνεται, νομίζω ότι προσπαθούμε να τραγωνίσουμε τον κύκλο σήμερα. Θα πρέπει να κάνουμε επιλογές δραματικές, δραστικές. Δηλαδή, στην Ήπεθρο ε, εστιάζουμε εκεί και έχουμε λιγότερα για τη Γεωργία. Αν δούμε τι μας μένει για τη Γεωργία. Καταρχάς, υπάρχει αυτό που αφορά χώρες ε, και περιοχές ε, μειονεκτούσες. Είναι εκ των όνων κάνευ και που σε σμένα κράτη είναι μεγάλος ο προϋπολογισμός αυτός, μεγάλα τα ποσά αυτά. Υπάρχει μετά το πρασίνισμα ή τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Αυτά τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Βλέπουμε το υπερβάλλον περιβαλλοντικό κόστος και αυτά τα μέτρα Ποιους αφορούν. Όλους τους γεωργούς. Ναι. Άρα και τους γεωργούς που θα χρειαστούν οικονομική στήριξη, που μας να τη βάλουμε όμως την ε, δεύτερη, στο δεύτερο πυλώνα. Γιατί ένας παραγωγός φρούτων, ας πούμε, ο οποίος ε, έβαλε χόρτο, ας πούμε, κάτω από τα, από τα φρούτα του, ε, δεν έχει δικαίωμα να ασφαλίσει, ας πούμε, το περιβόλι του κατά του χαλαζιού. Υπάρχει ένα μπέρδεμα με τους ε, στόχους. Θέλω να αναφερθώ σε κάτι που δεν αναφέρθηκε πολύ. Μας προτείνουν να βάλουμε στο δεύτερο πυλώνα επιστώσεις για τη διαχείριση των κρίσεων μέσω των οργανώσεων των παραγωγών, οι οποίοι θα μπορούσαν να βάλουν σε αποθεματικό κάποια χρήματα και αυτά, αυτά τα αποθεματικά αναδιανύμονται στους γεωργούς και εποφελούνται από μία πρικοδότηση που α, αυξάνουν το αποθεματικό κατά 65%. Η συζήτηση μας γίνεται παλαβή. Ο Άλμπερτ είπε ότι όλες οι χώρες δεν έχουν τις ίδιες επιλογές. Θα πρέπει πολύ γρήγορα στις προ... τις προτάσεις της Επιτροπής Γεωργίας να δούμε τι ακριβώς προτείνουμε. Γιατί νομίζουμε ότι προτείνουμε πράγματα, προτείνουμε τα πάντα στους γεωργούς. Αλλά κοιτάξτε, πάρτε λιγάκι ένα κομπιουτεράκι και δείτε ότι δεν γίνονται τα πάντα. Δεν μπορούμε να τα χώσουμε όλα στο δεύτερο πυλώνα. Ευχαριστώ, Κλάς και Ρίτα Έμερς. Η κυρία Κλάς. Παρακολούθησα προσεκτικά και διαπίστωσα ότι στο ερώτημα τι σημαίνει ανάπτυξη της υπαίθρου απαντούν πολύ διαφορετικά και ακόμα δεν είναι ξεκαθαρά τα πράγματα. Η ερώτησή μου έχει ως εξή. Τι εννοούμε πολυλειτουργική γεωργία για μένα δεν σημαίνει αναδρομή στο παρελθόν από μια εξειδικευμένη γεωργία, γεωργία να ξαναγυρίσουμε στην εκμετάλλευση με την αγρότησα να ψήνει ψωμί και γύρω να κυκλοφορούν οι γελάδες, τα γουρούνια και οι πάπιες. Χρειαστήκαμε πολλές δεκαετίες μέχρι να ξεσυνηθίσει να ψήνει ψωμί η αγρότησα γιατί δεν αξίζει τον κόπο και γιατί δεν είναι αρκετά στραμμένο προς το μέλλον. Νομίζω ότι πρέπει να αναζητηθούν και άλλοι πόροι εισοδήματος και τα όρια είναι ρευστά γι' αυτό. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να οριστεί αυτό το δεύτερο σκέλος της Γεωργίας. Αυτό μπορεί να ενταχθεί στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά μπορεί, αλλά μπορεί επίσης να είναι και τουρισμός, μπορεί να είναι, ε, όπως αλέχθηκε προηγουμένως, να βοηθήσουν οι νέες οδοί επικοινωνίας, το ταχύ διαδίκτυο, δεν υπάρχει περιορισμός εδώ. Αυτό που πρέπει να ε, προωθήσουμε ως ε, επικοινωνία είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή στην ουσία επιθυμούμε να εξυπηρετήσουμε, να στηρίξουμε την ύπεθρο, τις αγροτικές δομές και προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε και στο μέλλον αγροτικές περιοχές όπου υπάρχουν πολλές και καλές εκμεταλλεύσεις, αυτές είναι που είναι και πιο ισχυρές περιφέρειες. Για την ώρα δυστυχώς πολλά ε, πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή υπάρχουν πολλές στοχές αγροτικές περιοχές. Μια ερώτηση ωστόσο, δηλαδή δεν άκουσα καθόλου περί γυναικών. Πώς εντάσσονται εδώ οι γυναίκες, οι διάφορες ε, ενεργές αγρότησες. Δεν μπορούμε να τις λησμονήσουμε αυτές και θα πρέπει να είναι δυνατόν οι οργανώσεις αυτές να αναπτύξουν και δικές τους αυτόνομες ιδέες και να υλοποιήσουν προγράμματα. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και δεν επιτρέπεται να μείνει εκτός παρενθέσεως σε αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης Ευχαριστώ. Ρίτα. Κάθε φορά που μιλώ για θέματα υπαίθρου θέτω ένα ερώτημα με ποιον τρόπο θα βρούμε με ποιον τρόπο μάλλον θα βρούμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικότερα τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μήπως είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε κάποια κυκλικά ταμεία έτσι ώστε να μπορούν να συλλέγονται και χρήματα. Δεν είναι ανάγκη κάθε φορά να δαπανώνται όλα τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε, όλα τα κονδύλια τα οποία διαθέτουμε. Αν είναι δυνατόν να γίνει κάποια αποταμίευση ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν. Εσείς και καθηγητά τι γνώμη Δηλαδή, ε, κονδύλια να δοθούν και υπό την μορφή πιστώσεων, με υπολογισμό βεβαίως και των ενδεχομένων ε, αδυναμιών να αποπληρωθούν σε ορισμένε περιπτώσεις κτλ. Αλλά να το εξετάσουμε το όλον αυτό και από την χρηματοδοτική σκοπιά, διότι στο προσεχές μέλλον θα αισθανθούμε όλοι σημαντική πίεση, όχι μόνο στον αγροτικό προϋπολογισμό. Γνωρίζουμε ήδη πόσο πια σφιχτές θα είναι οι χώρες μέλη από εδώ και, και μπρος, στο μέλλον, πόσο δηλαδή περιορισμένα θα είναι τα χρηματοδοτικά τους περιθώρια. Αυτά λοιπόν που μπορούμε να, δω, να διαθέσουμε, πώς να διαθέσουμε με αποτελεσματικότερο τρόπο. Ευχαριστώ Μπριτά. Ο, καθηγητό, ο καθηγητής Βάντεν Πλούχ, όπως ε, είδατε η ε, παρέμβασή σας προκάλεσε πάρα πολλές ερωτήσεις, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και παρα, θα, θα, ε, θα με επιτρέψει να πω ότι είναι σημαντικό να μας βοηθήσετε να αντιληφθούμε καλά τη λειτουργία των μηχανισμών διαχείρισης του κινδύνου. Είτε πρόκειται για ε, συλλογική διαχείριση, είτε πρόκειται για ε, ατομική διαχείριση του κινδύνου. Μπορείτε λοιπόν να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε ακριβέστερα το τι πρέπει να κάνουμε και στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω όχι με τη σειρά που τέθηκαν. Να απαντήσω καταρχάς στο βασικό ερώτημα. Ποια είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου. Είναι απλό. Η ανάπτυξη της υπαίθρου στοχεύει στην ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και στη δημιουργία εδαφικής συνοχής κατά πρώτο λόγο. Κατά δεύτερο λόγο στοχεύει να στηρίξει ε, τη δημιουργία μιας νέας αγροτικής δραστηριότητας εξασφαλίζοντας την επάρκεια και την ασφάλεια των τροφίμων σε όλη την Ευρώπη. Και τρίτον βελτιώνει την ποιότητα ζωής στην υπαίθρο, στις αγροτικές περιοχές. Περί αυτού πρόκειται, έτσι αλληλοσυνδέονται η αγροτική δραστηριότητα και η ύπεθρος. Η ανάπτυξη της ε, γεωργικής δραστηριότητας και η ποιότητα ε, της ύπεθρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Εκεί όπου δεν ε, διεξάγεται αγροτική δραστηριότητα δεν έχει νόημα να μιλούμε για ανάπτυξη της ύπεθρου. Και από την άλλη, όταν έχουμε ε, αγροτική δραστηριότητα σε περιοχές, περιοχές κατεστραμμένες, ειδικά ε, πολύ έντονα εκπιομηχανισμένες, ε, εκεί δεν έχει νόημα πάλι η συζήτηση. Μιλούμε δηλαδή για την αμοιβαία εμβάθυνση, στήριξη του αγροτικού στοιχείου και του στοιχείου της υπαίθρου, της εξοχής από την άλλη. Αν είχαμε μόνο τις αγορές, και μάλιστα τις διεθνοποιημένες αγορές ε, σήμερα, ε, θα είχαμε μόνο ε, διακυμάνσεις πολύ υψηλές στις τιμές, ευμετάβολες καταστάσεις, αγρότες αμέσως θα εγκαθίστανται σε βόρειες περιοχές της Ευρώπης και θα εξαφανιζόταν η αγροτική δραστηριότητα στα ανατολικά και στο νότο της Ευρώπης, ε, αν μόνο οι αγορές δρούσαν ελεύθερα. Κανείς δεν το θέλει αυτό και γι' αυτό μας χρειάζεται πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου, παρόλο που είναι δύσκολο να δοθεί επαρκής ορισμός. Αυτό καταρχάς. Και βεβαίως Αυτά μας οδηγούν στην πολυλειτουργική ε, χρήση, στις πολυλειτουργικές χρήσεις γης και αυτά μας οδηγούν στην απάντηση ε, στο εξής ερώτημα. Γιατί χρειαζόμαστε χρήματα για την ανάπτυξη του υπαίθρου. Για να έχουμε μια πιο ελκυστική Ευρώπη, περισσότερο ισορροπημένη Μία ε, δραστηριότητα η οποία δεν θα εξαλειφθεί ξαφνικά εάν αφήσουμε τις αγορές να τα ρυθμίσουν όλα. Τώρα, μιλήσατε για τα ορυκτά καύσιμα. Συμφωνώ απολύτως και διαβάζοντας ένα από τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με χαρά είδα ότι το Κοινοβούλιο ενθαρρύνει το θέμα της ενεργειακής αυτάρκειας ε, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Αυτό μπορεί να γίνει και θα πρέπει να καταστεί σαφές την πρόταση για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Άρα πρέπει να έχουμε ψηλότερα επίπεδα στήριξης για να δώσουμε ενθάρρυνση κίνητρο στους αγρότες να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλήσαμε επίσης και για τη διαχείριση του κινδύνου. Συμφωνώ με την άποψη που εκφράσατε ότι δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα να ιδιωτικοποιούνται τα κέρδη και να κοινωνικοποιούνται τα, ε, οι κίνδυνοι και οι δυσμένειες. Αυτό ε, δεχομένω ε, θα οδηγούσε σε πολύ αρνητικές εξελίξεις τις οποίες δεν επιθυμούμε και των οποίων το τίμημα θα κληθούμε να καταβάλουμε σε μεταγενέστερο χρόνο. Και στην δική μου εργασία, την ερευνητική, έχω περιλάβει πολλές παραπομπές στη βιβλιογραφία και πολλές αναφορές για το θέμα αυτό. Τώρα, Εάν μπει ε, το πρασίνισμα θα πρέπει να μπει στο πυλώνα 1, να μην πάρει περισσότερα χρήματα ο πυλώνας αλλά να πούμε ότι το ποσό που κατά αποκοπή λαμβάνεται ανά εκτάρια θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε ως πληρωμή για ασφάλιση μέσω ασφαλιστικών προγραμμάτων ή μπορείτε να, το, να κάνετε αυτασφάλιση με συμπτώσεις να ασχοληθείτε εσείς προσωπικά για να έχετε κάλυψη στο μέλλον όταν οι αγορές θα λειτουργήσουν με αρνητικό τρόπο. Επομένως αυτό το θέμα των ασφαλιών δεν χρειάζεται να μπει ε, στον πυλώνα 2. Τώρα το πρασίνισμα. Ε, ένα θέμα που συζητείται ευρέω στην Ευρώπη. Δεν θα ήθελα αυτό το στοιχείο ε, να το περιορίσω σε έναν από τους δύο πυλώνες. Στην ερευνητική μου εργασία έχω περιλάβει πολλές ε, αγρονομικές γεωπονικές λεπτομέρειες. Μπορεί αυτό το στοιχείο να αξιοποιηθεί για να διαμορφωθούν οικολογικά, οικολογικά στοιχεία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες έτσι θα ενισχυθούν και θα μειώσουν πολύ το κόστος των ζυζανιοκτώνων φυτοφαρμάκων ε, που χρησιμοποιούν άρα θα είναι λιγότερο εξαρτώμενες αυτές οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Θα ήταν ε, πολύ έξυπνο να ε, κάνουμε το πρασίνισμα υποχρεωτικό και να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε την υιοθέτησή του παντού. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ο συνδυασμός αυτός. Και μάλιστα το πρασίνισμα μπορούμε να το πουλήσουμε με πολύ σημαντικό τρόπο, να το, κατα... να το καταστήσουμε πολύ ελκυστικό ε, στους Ευρωπαίους. Αν έχουμε π.χ. ισορροπημένη ε, βόσκηση στην κτηνοτροφική δραστηριότητα αλλάζουμε τη σχέση ε, κατανάλωσης καυσίμων και ε, παραγωγής κοπριάς η οποία χρησιμεύει ως λίπασμα. Επομένως, ανά 10 εκτάρια περιοχής ε, όπου έχουμε βόσκηση μπορούμε να, έχουμε λίπασμα και παραγωγή λιπάσματος το οποίο να αντιστοιχεί σε μετριασμό, σε απάλυνση ε, των ε, προβλημάτων των περιβαλλοντικών που να αντιστοιχούν σε ικανό αριθμό εκταρίων δασών που εξαφανίζονται λόγω των κλιματολογικών αλλαγών. Πρέπει γενικότερα να αλλάξουμε το σύστημα που προσφέρουμε. Ε, σήμερα η Ευρώπη λέει σε κάθε αγρότη ξεχωριστά αυτό μπορείς να κάνεις, αυτό δεν μπορείς, αυτό απαγορεύεται κτλ. Ένα γενικότερο, αυτά τα γενικά προγράμματα δεν λειτουργούν παντού. Μπορούμε να πούμε στις ομάδες παραγωγός παραγωγών. Εσείς υποβάλλετε μια πρόταση να μας πείτε πόσο θα συμβάλλετε στο μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της αλλαγής του κλίματος, πόσο, σε τι βαθμό θα καταστήσετε πιο ελκυστική την περιοχή σας, ε, πώς ακριβώς έχετε σκεφτεί δηλαδή να λειτουργήσετε και αν τελικά δεν ε, παρουσιάσετε τα ε, προϊόντα της δουλειάς σας, αν τελικά δεν καταφέρετε να επιτύχετε αυτά που έχετε πει, τότε θα σταματήσει η ενίσχυση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πιο ελκυστικό και έτσι θα μειώνεται και η γραφειοκρατία. Ω προ του νέου αγρότε, συμφωνώ απολύτω. Για να έχει ακόμα περισσότερη νομιμότητα δημοκρατική νομότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα θα πρέπει να δίνει περισσότερες απαντήσεις στην ανεργία των νέων, ε, θα πρέπει να βοηθά τους νέους ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση σε εκτάσεις και να έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μια ε, γεωργική δραστηριότητα. Το σημαντικό είναι να μην επινοήσουμε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά να ενισχύσουμε τη διασύνδεση ε, των υφιστάμενων μηχανισμών σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στην Ιταλία υπάρχει ένα πρόγραμμα διάθεσης δημοσίων γεών στους νέους προκειμένου να καλλιεργήσουν. Στη Γαλλία έχουμε ε, το Terre des ε, τις, ε, τα εδάφη σύνδεσης. Εκεί μπορεί να έχουν πρόσβαση οι νέοι και να ξεκινήσουν γεωργική δραστηριότητα. Στις κάτω χώρες έχουμε παρεφερεί συστήματα. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε αυτούς τους τοπικούς, τους εθνικούς μάλλον μηχανισμούς για να μειωθεί η γραφειοκρατία και έτσι και για να καταστεί πολύ πιο αποτελεσματική πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Τώρα, υπάρχει ε, για τους ε, τέσσερις άξονες. Πράγματι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να αποδυναμωθεί το περιεχόμενο και γίνεται λόγος για την καινοτομία η οποία ενίοτε κυριαρχεί. Αν όμως μελετήσατε προσεκτικά την πρόταση θα δείτε τα εξής. Προβάλλεται το εξής επιχείρημα. Ε, στην επτατή περίοδο τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα είναι ίσα ή λιγότερα με ό,τι έχει ήδη γίνει την προηγούμενη επτατή περίοδο. Επίσης σε επίπεδο του ε, leader ε, ε, προβάλλεται το επιχείρημα ότι οι προηγούμενε προσπάθειε θα πρέπει να συνεχιστούν. Αν τα πάρουμε όλα αυτά σοβαρά υπόψη, τότε έχουμε χτίσει ένα ε, επαρκέ αμυντικό τείχο, επιτρέποντα παράλληλα περισσότερη ευελιξία. Από εκεί και πέρα, τι άλλο έχω σημειώσει. Το θέμα τη υψηλή τεχνολογία και του χαμηλού κόστου. αγροτική εκμετάλλευση υψηλή τεχνολογία και αγροτική εκμετάλλευση χαμηλού κόστου. σύγκριση μεταξύ των δύο δεν είναι πολύ χρήσιμο εγώ ή εσείς ή πτώση εμείς να αποφασίσουμε ποιο, ποια είναι η καλύτερη άγουσα. Η, η κατάσταση στην αγορά το αποφασίζει αυτό και έχει αλλάξει άρδιν η κατάσταση στην αγορά. Οι νικητές, οι καλύτεροι μαθητές των αγροτικών εκμεταλλεύσεων υψηλής τεχνολογίας που ήταν το μότο του παρελθόντος δεν είναι καθόλου νικητές σήμερα που έχουν αλλάξει οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Σήμερα νέοι μπαίνουν στα αγροκτήματα, τα αλλάζουν, λαμβάνουν αποφάσεις. Επομένως η αγροτική εκμετάλλευση χαμηλού κόστους είναι πιο βιώσιμη και είναι και πιο διαφοροποιημένη έχει πιο ευρία γάμα δραστηριοτήτων, πόσο μάλλον να είναι πολυλειτουργική. Έτσι αυτό ε, είναι πολύ ελκυστικό για τους νέους. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι εμπειρικές μελέτες. μελέτες. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι επειδή το λέω εγώ, αλλά το έχουμε δει στην πράξη. Ε, όλο και περισσότεροι άνθρωποι πείθονται από αυτού του είδους την ε, πολυλειτουργική γεωργική δραστηριότητα. Και τέλος, δύο λόγια για το μέλλον. δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις πληρωμές αναχώρα ε, βάσει ε, των νεκταρίων. Επομένως, για να... Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ερευνηθεί το έδαφος πάνω στο οποίο θα στηριχθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να τα εξετάσουμε από κοινού με τους στόχους. Ίσως θα παραμείνουν οι διαφορές και καλό θα ήταν να έχουμε καλύτερη δυναμική και όχι επιβολή άνωθεν των μέτρων. Να δούμε την ανάπτυξη της υπαίθρου ως μια διαδικασία διαπραγμάτευσης οι ομάδε παραγωγών να υποβάλουν τι προτάσει του, να λένε ότι εμεί αυτά μπορούμε να κάνουμε, αυτά μπορούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία, στι ε, ε, επίσημε τοπικέ αρχέ και σε ποιο βαθμό μπορείτε εσεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση να μα βοηθήσετε. Τι είδου χρηματοδότηση ε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε εμεί οι ομάδε παραγωγών. Και μετά μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτο να έχει ένα απλό σύστημα ελέγχου, αλλά αξιόπιστου ελέγχου, να έχει μια πολυλειτουργική προσέγγιση και να απαντάει, να ανταποκρίνεται σε αυτά τα αιτήματα. Νομίζω ότι αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουμε και σας εύχομαι ε, σε εσάς που είστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλή δύναμη στη διαδικασία της ε, συναπόφασης προς αυτή την κατεύθυνση. Και μία ε, τελευταία παρατήρηση έχω να κάνω κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να παρακολουθήσω τη συζήτηση, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να χάσω την πτήση μου και πρέπει σε πέντε λεπτά να φύγω. Λυπούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ευχαριστούμε τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Βαγγενίκεν. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση στα πλαίσια του εργαστηρίου που είχαμε. Χαιρετίζουμε λοιπόν, αποχαιρετούμε τον καθηγητή και πάμε στο σημείο 6 μερισίας διάταξης ή μάλλον στο σημείο 5 διορθώνει ο πρόεδρο, στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων. Η συγγήτρια Μάρι Πόλσεν θα κάνει μια ανταλλαγή απόψεων για αυτή τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προστασία και την ευμερία των ζώων. Έχουμε το άρθρο 13 της συνθήκης, αφορά, για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζει ότι τα ζώα είναι αισθανόμενα όντα και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ευημερία των ζώων κατά, την εφαρμογή και την, κατά τη διατύπωση και την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών. Η ε, Κομισιόν στις 19 Ιανουαρίου ε, υιοθέτησε μια στρατηγική για την προστασία και την ευημερία των ζώων και η Αντιπρόεδρος, η κυρία Πόλσεν, είναι ε, η συντάκτρια αυτής της γνωμοδότησης πρωτοβουλίας, την οποία θα παρουσιάσει. Της δίνω το λόγο. Μάριτ, έχεις το λόγο έχουμε να εξετάσουμε αυτή την ε, ε, έκθεση στις 19 και 20 Μαρτίου και στις 30 Μαρτίου ε, θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Μάρι, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Η πρόταση της Κομισιόν βασίζεται στην έκθεση πρωτοβουλίας που το Κοινοβούλιο και ειδικά η Επιτροπή μας ε, είχε ψηφίσει την Άνοιξη του 2010. Έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε, να απλουστεύσουμε και να διευκρινίσουμε τα θέματα που αφορούν την ευημερία των ζώων. Το κείμενο μπορώ να πω ότι είναι αρκετά αόριστο δεν είναι πολύ σαφές. Και πριν από δύο χρόνια είχαμε πει ότι χρειαζόμαστε κάποια πράγματα. Έχουμε ορισμένε απαιτήσει, αλλά οι οποίες δεν εμφανίζονται ή αποδυναμώνονται στο κείμενο. θα πρέπει να προωθούμε την ευμερία των ζώων ε, με βάση τα όσα προβλέπουν οι συνθήκε. Άρθρο 13, τι συνθήκε για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε μεγάλο περιθώριο ευελιξία. Εδώ πρέπει να καλύψουμε όλα τα ζώα, εκτό από τα άγρια ζώα. Δηλαδή, όλα τα ζώα με τα οποία έρχεται σε επαφή ο άνθρωπος ή με τα οποία ασχολείται ο άνθρωπος. Μην ξεχνάμε επίσης ότι έχουμε κοινέ αρρώστιες κατά το 70% με τα ζώα. Ε, το 95% όλων των ζώων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης είναι ζώα που τα χειρίζονται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, που έχουν την ευθύνη για αυτά. Ε, οι άνθρωποι ζουν με τα ζώα και ζουν και χάρη στα ζώα. Θέλω να περιοριστώ στα ζώα της εκμετάλλευσης κυρίω στις δυνατότητες που υπάρχουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι Παύλα Γεωργοί. Αν λάβουμε υπόψη μας τη σημερινή κατάσταση και το έγγραφο που θα δώσουμε προς μετάφραση αύριο, λέει, έχει 23 αναφορές στους διάφορους κανόνες, οδηγίες, κανονισμού. που σήμερα αφορούν τους γεωργούς και τα ζώα τους. Έχουμε 27 κράτη-μέλη με διαφορετικούς κανόνες, διαφορετικούς ελέγχους σε διάφορα επίπεδα. Το πρόβλημα του σεβασμού των κανόνων είναι ένα δεδομένο. Επίσης, το πρόβλημα της κατανόησης. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην Ευρώπη σήμερα. Έχουμε ας πούμε τη, τις α, κότες Ένα πρόβλημα για το οποίο έχουμε μιλήσει εκατοντάδες φορές. Σήμερα είναι σαν να τιμωρούμε αυτούς που σέβονται τους κανόνες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με κανόνες όπως αυτούς που έχουμε σήμερα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τους παρακάμψουμε σε τόσες πολλές χώρες. Ε, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συνεχιστεί, ενώ σε άλλες χώρες οι γεωργοί είναι υποχρεωμένοι να σέβονται αυτούς τους κανόνες υπέρ των ζώων. Αυτό το πράγμα, αυτή η διαφορά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Επίσης, υπάρχει μια οδηγία που θα εφαρμοστεί το Φεβρουάριο του 2013 για, τα, για τους χείρους. Και ξέρουμε ότι θα υπάρξουν, ήδη από τώρα το ξέρουμε, ότι θα υπάρξουν ε, πολλά κρατημέλη που είναι αδύνατο να μπορέσουν να σεβαστούν μέχρι τότε τους κανόνες. Σκεφτείτε λιγάκι το θέμα του σεβασμού των κανόνων που υπάρχουν. Στις ε, σκανδιναβικές χώρες ε, έγινε μία εκστρατεία την περασμένη εβδομάδα, όπου είπαμε μέσα από την εκστρατεία ότι δεν πρέπει να αγοράζουμε βόλιο κρέας. Όχι, εγωπρόβιο κρέας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ε, σκοτώνουμε αυτά τα ζώα χωρίς να τα υπνώσουμε πριν. Χωρίς να τα κοιμήσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μία παραποίηση, μία χειραγώγηση των πληροφοριών ε, υπάρχουν ας πούμε κάποιες ε, μειονότητες, μια θρησκευτική μειονότητα η οποία έχει διαφορετικούς κανόνες ε, σφαγής των ζώων ας πούμε. Ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με, όλες, όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Η κατάσταση είναι χαόδης. Και, και είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Γιατί τελικά ποια είναι, ποιος είναι ο ορισμός της ευημερίας του, των ζώων. Γιατί είναι τόσο δύσκολος αυτός ο ορισμός σήμερα. Γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εγώ ήρθα σε επαφή με όλες τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις, οργανώσεις ε, αγροτών, οργανώσεις ε, προστασίας του περιβάλλοντος, με επιστήμονες, με εκπροσώπους ε, σφαγίων, με κτηνιάτρους. Άκουσα όλους. Και μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις παρουσιάζω ε, αυτή την πρόταση, η οποία θα μεταφραστεί αύριο. Η ιδέα μου είναι να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μία απλούστευση, σε μία απλή νομοθεσία, σαφή, εναργή, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και είναι και πρακτική. Γιατί δεν μπορούμε έτσι να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε κανόνες, να φτιάχνουμε νομοθετήματα, τα οποία είναι απλώς ε, φλιναθήματα και που δεν λειτουργούν όμως ε, στην πράξη, δεν λειτουργούν στην καθημερινότητα. Επομένως, εγώ αυτό θα, θα ήθελα να ζητήσω είναι ένα νόμο πλαίσιο. Κοινούς κανόνες. Όπως παραδείγματος χάρη έχουμε για τα τρόφιμα. Πριν από 12 χρόνια εγώ συμμετείχα σε αυτή την ε, σύνταξη των κοινών κανόνων για τα τρόφιμα και θυμάμαι ότι πάρα πολλοί ήταν ε, πεπισμένοι ότι αποκλείεται να λειτουργούσε το όλο σύστημα αυτό. Γιατί υπήρχαν τόσο πολλές διαφορές μεταξύ των 15 τότε που ήταν αδύνατον να λειτουργήσει το σύστημα. Οι διαφορές όντω ήταν τεράστιες και δεν φανταζόμαστε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα νόμο πλαίσιο, για να το πω έτσι. Αλλά σήμερα τα έχουμε καταφέρει, έχουμε ένα πλαίσιο. Φυσικά ένα τέτοιο, ένα τέτοιο νομοθέτημα δεν, έχει όλες, δεν μπαίνει σε όλε τι λεπτομέρειε. Και το Common Food Law δεν μπαίνει σε υπερβολικές λεπτομέρειες. Απλώς είναι ένα νομοθέτημα πάνω στο οποίο βασίζονται όλες οι υπόλοιπε ειδικέ νομοθεσίες, όλα τα υπόλοιπα νομοθετήματα, οδηγίες, κανονισμοί κτλ. Θα ήθελα παραδείγματο χάρη να έχω έναν ορισμό για του γάμματα φόμικρον Κάτι που να είναι εύκολο, κατανοητό. και να ισχύει παγκόσμια. Γιατί αν έχουμε τέτοιους σαφείς κανόνες θα μπορούμε και στις ε, διμερείς συμφωνίες και στις πολυμερείς συμφωνίες να πούμε αυτό είναι ο κανόνας και σεβόμαστε τον κανόνα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, του ΟΙΤΕ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πρέπει να υπάρχει και δίκαιος ανταγωνισμός. Δεν μπορούν να υπάρχουν τόσες διαφορές στην ενιαία αγορά. Αυτό, άλλωστε, είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που θα πρέπει να την ύπαρξή τους να θυμόμαστε πάντοτε στη Γεωργία. Δηλαδή, μιλώ για τον έντιμο ανταγωνισμό. Από την εμπειρία της ζωής μου και επειδή είμαι και σε κάπως προχωρημένη ηλικία έχω συναντήσει και γνωρίσει πάρα πολλούς αγρότες σε πολλές χώρες του κόσμου και ήμουν και δημοσιογράφος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγροτική οικονομία. Αυτή λοιπόν η εμπειρία ζωής μου δείχνει ότι δεν υπάρχει σχεδόν κανένας αγρότης που να μην αγαπά τα ζώα του. Οι αγρότες ζουν κοντά στα ζώα, μαζί με τα ζώα και ζουν από τα ζώα. Τα υγιή και ήρεμα ικανοποιημένα ζώα είναι πολύ πιο εύκολο να ε, ζήσει μαζί τους και να τα εκμεταλλευτεί με τον σωστό τρόπο από ε, ζώα τα οποία είναι ενδεχομένως ε, ασθενή ή σε κακή κατάσταση. Αυτά λοιπόν θα ήθελα τώρα να μάθω και από εσάς τι θεωρείτε ότι είναι σημαντικό για την προστασία των ζώων. Η προσπάθεια αυτή έχει αρχίσει εδώ και μια δεκαετία με προσπάθειες άλλων συναδέλφων και εγώ θέλω να συνοψίσω ξανά ότι θα πρέπει να είναι ένας ορισμός σαφής και εύκολο να ε, μεταφερθεί, να καταστεί γνωστό. Ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο, την κυρία Πόλσεν. Ε, θέλουν πολύ να συμμετάσχουν στη συζήτηση, μην ξεχνάμε και το χρόνο, γιατί έχουμε και τη συνεδρία των συντονιστών με, την, ε, με τα κοινοβούλια των βαλτικών χωρών. Η κυρία Νταντσίλα είναι η πρώτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, εκ μέρους του Ντασιάν Σέρμπου, που είναι ε, συντονιστής εκ μέρους των σοσιαλιστών. Πιστεύουμε ότι οι γεωργοί θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την ευημερία των ζώων και να ανταμείβονται οικονομικά για αυτή την προσπάθεια. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα να δίνουν χρηματοδότηση από το δεύτερο πυλώνα σε νέες γεωργικές πολιτικές που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την ευημερία των ζώων ταυτόχρονα. Η στρατηγική για την ευμερία των ζώων μέχρι το 2015 θα πρέπει να λαμβάνει ε, υπόψη ε, ιδίως το πρόβλημα των αδέσποτων ε, σκύλων. Η στρατηγική θα πρέπει να απαιτεί από τον κόσμο να δρά με υπευθυνότητα απέναντι στα οικόσιτα ζώα, ούτως ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο του πολλαπλασιασμού των αδέσποτων ζώων και σκύλων ιδιαίτερα. Για να βελτιώσουμε την ευημερία των ζώων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, του κάθε κράτους μέλους και θα πρέπει να προβλέψουμε μεταβατικές περιόδους, ούτως ώστε να επιτύχουμε την εναρμόνιση που είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η σκιώδη συγγήτρια του Λαϊκού Κόμματος είναι η κυρία Γέγκελ. Θα ήθελα να την εκπροσωπήσω και παίρνω το λόγο για να σας πω ότι η ενίσχυση των κοινοτικών νομοθετημάτων με ένα ε, νέο ε, νομοθετικό πλαίσιο από το 2014 είναι πάρα πολύ σημαντικό κυρίως ε, και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα στα χειροστάσια. Ε, δεν θέλουμε να υπάρξουν ανισορροπίες. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο κάποιους έναντι κάποιων άλλων για τα εγωπρόβατα. Σε ορισμένους υπάρχουν, ε, εφαρμόζονται κάποιοι κανόνες, άλλοι δεν ε, πρέπει να σεβαστούν αυτούς τους κανόνες. Θα πρέπει να πλουστεύσουμε όλα αυτά τα πράγματα η απλούστευση είναι πάντα καλό πράγμα. Και θα πρέπει να έχουμε κάποια απλά κριτήρια με δείκτες επιστημονικούς που προτείνονται από τους ειδικού. Εμείς δεν είμαστε εμπειρογνώμονες στην ε, κτηνοτροφία. Οι κτηνίατροι θα πρέπει να μας δώσουν κάποια στοιχεία που να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, ε, ούτως ώστε να προωθήσουμε και την ανταγωνιστικότητα για τους κτηνοτρόφους με σεβασμό της ευημερία των ζώων. Ε, Λαμβάνοντα υπόψη κάθε ειδικό τομέα. Γιατί οι, κτηνοτρόφοι μας, κτηνίατροι μα λένε ότι δεν είναι ίδιες ανάγκε παντού α, σε όλα τα είδη ζώων. Επομένω, οπωσδήποτε θα πρέπει να δώσουμε τον λόγο στου ε, κτηνιάτρου, που είναι οι δήμονε. Επίση, ε, κάνουν μια απόπειρα σε Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγαλύτερη διαφάνεια. Καλό είναι αυτό. Επίση, κάτι άλλο σημαντικό είναι η ενημέρωση του καταναλωτή. Ακόμη και αν βάλουμε ετικέτε, ακόμη και αν κάνουμε σημαντικέ προσπάθειε. Αν ε, δεν εξηγήσουμε στου καταναλωτέ ότι η ευημερία των ζώων είναι προστιθέμενη αξία, αποτελεί προστιθέμενη αξία, ε, τη στιγμή τη αγορά ο καταναλωτή αυτό το πράγμα δεν θα το λαμβάνει υπόψη καθόλου. Είναι πολύ σημαντικό επίση να εφαρμόσουμε όλα όσα υπάρχουν σε νομοθετικό επίπεδο, γιατί δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, Γιατί τι νόημα έχει να είμαστε πιο απαιτητικοί, αν σε μια χώρα χ, ας πούμε, δεν σεβόμαστε τίποτα. Ε, και τη σεβόμαστε, ας πούμε, σε σεβόμαστε τους κανόνες ε, σε μια άλλη χώρα. Λέει, το θέμα του σεβασμού των κανόνων με τον ίδιο τρόπο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, αφού εφαρμοστούν οι κανόνες, μετά θα πρέπει να ανεβάσουμε τον πύχη. Ε, επίσης, ε, ενημέρωση μέσω της ετικέτας, αλλά και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Δεν έχει κανένα νόημα να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία στην ετικέτα, αν ο καταναλωτής δεν καταλαβαίνει τι νόημα έχει αυτό. Επίσης, υπάρχουν πολλές δεσμεύσεις, πολλές ρητορίε, ακούγονται πολλά λόγια, αλλά λίγα ε, συγκεκριμένα πράγματα, λίγα έργα. Οι παραγωγοί έχουν επενδύσει Η πρόταση της Κομισιόν ε, για τις επενδύσεις ε, απαιτούν ε, τεράστιες προσπάθειες από τους παραγωγούς, αλλά η χρηματοδότηση της Κομισιόν που προβλέπει η Κομισιόν είναι πάρα πολύ ανεπαρκής. Τι νόημα έχει να ζητάμε από τους εκμεταλλευτές να κάνουν πολλές προσπάθειες, αν και η Κομισιόν δεν προβλέπει μια κατάλληλη χρηματοδότηση. υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη χρηματοδότηση που προβλέπει η Κομισιόν. Θα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια και η Κομισιόν στις διεθνείς συμφωνίες για την ευμερία των ζώων, στις ε, διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει ε, και στις διμερείς συμφωνίες και στις συμφωνίες που ε, υπογράφονται σε επίπεδο ΠΟΕ, σε πολυμερές επίπεδο. Γιατί δεν είναι σωστό ηθικά και δεοντολογικά να ζητάμε από τους δικούς μας ε, γεωργούς και κτηνοτρόφους σε περίοδο κρίσης όλο και περισσότερα πράγματα και παράλληλα όταν υπογράφουμε συμφωνίες με τρί, τρίτες χώρες να κλείνουμε τα μάτια και να μην απαιτούμε τίποτα από αυτούς. Να μην απαιτούμε αυτά που απαιτούμε από τους δικούς μας ε, τους ε, γεωργούς και κτηνοτρόφους. η ευημερία των ζώων λοιπόν και ο σεβασμός αυτής από αυτούς είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σωστή η νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων και τα 150 εκατομμύρια ευρώ για την καλή διαβίωση των ζώων. Μέχρι τώρα η νομοθεσία βέβαια δεν ήταν συνεπής. Για παράδειγμα δεν υπάρχει ε, νομοθεσία σήμερα για τις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες και για τα ε, βοηθή που, προσδίδει την παραγωγή κρέατος. Το ίδιο δεν επιβάλλεται η ισχύουσα νομοθεσία και γι' αυτό είναι σημαντικό το νέο βήμα. Η έκθεση αυτή θα δώσει μια ένδειξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το τι επιθυμούμε να δούμε να συμβαίνει στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πόλσεν για την πολύ επικοδομητική διστάση ως εισηγήτριας. Είπε ότι ακούει τις απόψεις των άλλων πολιτικών ομάδων και νομίζω ότι σημειώθηκε και σημαντική συμφωνία στα σημαντικά θέματα. Για μας οι προτεραιότητες είναι ένα καλύτερο σύστημα επιβολής της νομοθεσίας με ορόσημα τα οποία θα επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώνει αν οι χώρες μέλη ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, διότι σήμερα χωρίς το σύστημα αυτό ε, τα πράγματα καθυστερούν πάρα πολύ. Και ο ίδιος ο κύριος Νταλή ε, ζήτησε, ε, αναγνώρισε την αξία του συστήματος αυτού όταν μίλησε στην ομάδα εργασίας για την καλή διαβίωση των ζώων. Και οι χώρες μέλη που δεν θα εφαρμόζουν την νομοθεσία έγκαιρα θα δέχονται κάποια βοήθεια για να επανέλθουν στην ορθή ε, οδό, ας το πω έτσι. Όπως είπαν και άλλοι και για τον δεύτερο πυλώνα, αλλά σημαντικό είναι επίσης να γίνει και εκπαίδευση του προσωπικού. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω των υφισταμένων θεσμών. Η ίδια υψηλά επίπεδα πρέπει να ισχύουν βέβαια και για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ίδια δηλαδή ε, πρότυπα που ισχύουν για τους δικούς μας Γιώργους, για παράδειγμα για τους δικούς μου στην Ουαλία που ευχαρίστως ε, εκπλούν τις υποχρεώσεις τους ό,τι αφορά την τήρηση υψηλών προδιαγραφών, αλλά το ίδιο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και για τις εισαγωγές από άλλα μέλη του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και η σωστή επισήμανση γιατί δεν θέλουμε να βρεθούν σε δυσμενή θέση οι παραγωγοί οι οποίοι σέβονται τα υψηλά πρότυπα. Νομίζω ότι υπάρχει καλή συνεργασία και χαίρομαι γι' αυτό για την έκθεση και έτσι με τον τρόπο αυτό θα δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ η κυρία Γέγκλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Πόλσεν για την πρώτη αυτή συζήτηση και νομίζω ότι μια πρώτη έκθεση, αυτή δηλαδή που περνά τώρα από τη μετάφραση, θα αντιλάβουμε και αυτήν. Εγώ είμαι βεβαία ότι εάν εξετάσουμε τα τελευταία δέκα χρόνια θα διαπιστώσουμε ότι έχουν γίνει βήματα και θα παρακαλέσω και τις και τους συναδέλφους να το δουν αυτό. Ιδιαίτερα για παράδειγμα για τον κανονισμό για τις οτόκους όρνηθες. Βλέπουμε βέβαια τις μεγάλες ελλείψεις που ωστόσο βασίζονται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε την ευκαιρία, δεν είχε τη δυνατότητα έγκαιρα και επαρκώς να συνεργαστεί και να παρέμβει στις χώρες μέλη. Να συνεργαστεί με τις χώρες μέλη και να παρέμβει σε αυτές όταν βλέπει ότι τα πράγματα δεν προχωρούν και δεν εφαρμόζονται σωστά. Αν θέλουμε πραγματική προστασία των ζώων θα πρέπει να καταθέσουμε μια έκθεση που να στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα σημαντικά ζητήματα και πρέπει να ορίσουμε κιόλα ποια είναι τα βασικά ζητήματα και αυτό μπορεί να γίνει βήμα-βήμα. Εγώ θεωρώ ότι ο αγρότης έχει κάθε συμφέρον να φροντίζει και να περιποιείται τα ζώα του, διότι με αυτά ε, κερδίζει τα προστοσύν και είναι πολύ καλύτερα να έχει στη διάθεσή του υγιή ζώα και όχι άρρωστα ή ε, καχεκτικά. Γι' αυτό και πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι ε, τελευταίες εξελίξεις ε, στη γνώση για την κτηνοτροφία. Πολλά πράγματα είναι διαρκώς ρευστά και αυτό που λένε βεβαίως οι Γεωργοί είναι ότι δεν θέλουμε και κάθε έξι μήνες ή κάθε λίγα χρόνια να δεχόμαστε νέους δεσμευτικούς κανόνες. Εγώ για παράδειγμα μου λέει ένας Γεωργός έχτισα τους τάβλους σύμφωνα με τους τότε ισχυούντες κανονισμούς και μάλιστα με ενίσχυση. Και τώρα ξαφνικά έρχονται και μου λένε όχι πρέπει να είναι διαφορετική η στάβλη αυτή. Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και σε αυτές τις ανησυχίες των γεωργών χωρίς να τους επιβαρύνουμε με υπερβολική γραφειοκρατία. Και ταυτόχρονα να πούμε ότι η προστασία των ζώων, η καλή διαβίωσή τους είναι σημαντική και για μας. Κατά την άποψή μου τα σημαντικότερα ζητήματα πρέπει να μας απασχολήσουν είναι η εφαρμογή πρώτα των υφιστάμενων νομοθετικών μέτρων. Επίσης η έγκαιρη προειδοποίηση και η έγκαιρη παρέμβαση. Τι το θέμα και ποιο νομοθετικό πλαίσιο θα ισχύει για την προστασία των ζώων. Θα υπάρξουν ειδικά νομοθετήματα, θα ενταχθούν στην ευρύτερη αυτή νομοθεσία και με ποιο τρόπο θα την αντιμετωπίσουμε. Το ερώτημα είναι και τι γίνεται επίσης με τις νομοθετικές πράξεις από τις οποίες ή μάλλον για τι οποίε αναμένουμε ότι θα έπρεπε να είχε εκδώσει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή υπάρχει χώρο εδώ για ειδικά ζητήματα. Αυτά πω θα ενταχθούν ή πώς θα υπαχθούν σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, ε, ε, επιστημονικά θεμελιωμένοι δείκτες που νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Από την άποψή μου είναι σημαντικό να πούμε ότι η πω θα υπαχθουν σε αυτο το νομοθετικο πλαισιο επισης επιστημονικα θεμελιωμενοι δεικτε που νομιζω οτι αποτελεί τη βάση. Δεν υπάρχει χώρος εδώ για ιδεολογίες. Πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι γραμμές και τότε μόνο μόνον θα έχουμε την υποστήριξη των ανθρώπων οι οποίοι ε, ενδιαφέρονται άμεσα. Κριτήρια επίσης τα οποία να γίνονται δεκτά και στις 27 χώρες μέλη και να μπορούν να εφαρμοστούν. Εν προκειμένου ίσως πρέπει να σκεφτούμε επίσης τι θα πρέπει να κάνουμε για να φέρουμε και τις 27 χώρες μέλη σε μία κοινή αφετηρία πριν αναπροχωρήσουμε στην επιβολή νέων προτύπων. Στην έκθεση αυτή θα πρέπει να κάνουμε και μια διασύνδεση και με τις μεταφορές των ζώων που και αυτές έχουν σχέση με την καλή διαβίωση των ζώων. Προδεκαετίας, κυρία Πόλσεν, θυμούμε ότι ήταν μέγα τότε το θέμα οι ικανότητες και οι γνώσεις των ανθρώπων που χειρίζονται τα ζώα. Είναι μόνο οι αγρότες, είναι και οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων που τα μεταφέρουν. Είναι θέμα αυτό και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Το τρίτο και τελευταίο και από τα πιο σημαντικά εμείς μπορεί να φτιάχνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι νομοθεσίες θέλουμε. Εάν ωστόσο δεν εξετάσουμε και τις διμερείς συμφωνίες που συνάπτουμε εάν ανταποκρίνονται στα πρότυπα αυτά, εν τέλει θα χάσουν το παιχνίδι η παραγωγή μας, διότι ο καταναλωτής εν τέλει θα αγοράσει αυτό που θεωρεί ότι είναι πιο συμφέρον για αυτόν. Ίσως εισαγωγέ από χώρε όπου οι, οι οργανώσει προστασία των ζώων δεν είναι τόσο ισχυρές όπως εδώ στην Ευρώπη. Θα χρειαστεί λοιπόν να εξετάσουμε ξανά και ξανά και να συζητήσουμε με όλους αυτούς που ασχολούνται με τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Αυτό για μένα είναι σημαντικότατο θέμα. Τότε μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί και να καθιδρύσουμε μια καλύτερη προστασία των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Πόλσεν, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είμαι βεβαίω ότι θα υποβληθούν πολλές τροπολογίες, αλλά πάλι επίσης είμαι βεβαίω ότι με τη συνεργασία μαζί σας θα καταλήξουμε σε καλούς συμβιβασμούς. Κύριος τώρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πόλτσον, μην ε, πάρετε τα σχόλιά μου προσωπικά, έτσι. Αλλά όντως, δεν ξέρω αν η λύση είναι περισσότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το θέμα είναι η εφαρμογή της. 27 κράτη-μέλη έχουμε με διαφορετική νοοτροπία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν εφαρμόζονται οι νόμοι αυτοί σε ορισμένα κράτη-μέλη. Έχουμε επαρκείς νόμους για την μεταφορά των ζώων, για την, ε, για την σωστή ρύθμιση και διαμόρφωση των ε, κλοβών ε, στα πουλερικά. Δεν εφαρμόζονται σωστά. Για ένα σωρό πράγματα έχουμε νόμους. Νομίζω και στοιχηματίζω ότι θα δούμε μια επανάληψη του ίδιου έργου. Και ε, υπησέρχεται εκεί πολιτική, το πολιτικό ορθό ε, ορισμένοι ε, σφαγιάζουν ζώα με πολύ άσχημη με άσχημο τρόπο και επειδή έχουμε, είμαστε δειλοί δεν θέλουμε να το στυλιτεύσουμε αυτό όπως θα έπρεπε. Έγιναν σχόλια για επιδοτήσεις ε, όμως είναι άδικο αυτό για τους αγρότες που έχουν δανειστεί για να συμμορφωθούν με τα ευρωπαϊκά προαπαιτούμενα. Ε, τελούν τώρα σε συγκριτικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Υπάρχει και το θέμα του ΠΟΕ. Δεν μπορεί να απαγορεύσει κανείς ε, την εισαγωγή κάποιου πράγματος επειδή διαφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο έχει παραχθεί αυτό το προϊόν. Ε, διαφορετική είναι η λύση. Η λύση είναι οι καταναλωτές να κάνουν αυτό ε, που έκαναν πριν από 30 χρόνια, όπου έλεγαν ότι θέλουμε αυγά ελευθέρας βοσκής. Λειτουργεί μόνο αυτό. Οι καταναλωτές είναι αυτοί που έχουν πυγμή και δύναμη και μπορούν να πούν στους, ε, στα σημεία λιανικής, στις μεγάλες επιχειρήσεις, τι είδους ε, κρέας θέλουν να καταναλώνουν. Είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η νοτροπία για την ε, καλή διαβίωση των ζώων. Στη χώρα μου έχουμε το RSPCA. Συμβάλλει οικονομικά ο κόσμος και η οργάνωση αυτή διώκει όσους παραβαίνουν εξετάζουν ε, την ε, καλή ή μη διαβίωση των ζώων, γίνονται αναφορές στην RSPCA και ε, ε, αναλαμβάνεται δράση. περισσότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν είναι λύση κατά την άποψή μου. Ευχαριστώ. Μην ξεχνάτε και το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητοί βουλευτές. Το λέω για τους υπόλοιπους ομιλητές. Ευχαριστώ. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τις αυστηρότερες προδιαγραφές προστασίας των ζώων από όλο τον κόσμο. Και αυτό μας καθιστά υπερήφανος. Από την άλλη πρέπει να οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι από αυτές τις αυστηρές προδιαγραφές προκαλούνται και ορισμένα προβλήματα. Και αυτό λέχθηκε ήδη, δηλαδή ότι άλλες χώρες δεν τηρούν τέτοιες αυστηρές προδιαγραφές. Άρα, εν τέλει, παράγουν φθηνότερα. Και αυτά τα φθηνότερα προϊόντα αγοράζονται τελικά ευχαρίστως από τους ευρωπαίου καταναλωτές οι οποίοι δεκάρα δεν δίνουν για το πώ παρήχθη το προϊόν. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να αγοράσουν με τα ίδια χρήματα περισσότερο προϊόν. Μπορούμε να πούμε χιλιάδες φορές εμείς ότι θα ήταν ευκταίο οι εισαγωγέ να περιορίζονται εφόσον δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές η Κομισιόν θα μας υπενθυμίσει ξανά και ξανά ότι στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τέτοια μέτρα. Ο ΠΟΕ δεν προβλέπει μέτρα που να επιτρέπουν την αναφορά σε προδιαγραφές προστασίας των ζώων για να περιοριστούν οι εισαγωγές. Εφόσον λοιπόν επιβάλλουμε νέα, τα νέα αυτά πρότυπα, θα αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των εισαγόμενων προϊόντων. Εξάλλου, πρέπει να μην λησμονούμε ότι η διαρκής αύξηση των τιμών των προϊόντων δυσαρεστεί τους καταναλωτές. στην Ευρώπη δεν εγκαταλείφθηκε η παραδοσιακή παραγωγή αυγών επειδή δεν ήταν αποδοτική, αλλά επειδή δεν, μάλλον δεν εγκαταλείφθηκε για τους λόγους, παρά επειδή δεν ήταν αποδοτική. Υπάρχει μεγάλο χάσμα με, ανάμεσα στα εισοδήματα των διαφόρων ε, στρωμάτων του πληθυσμού. αυτοί που ζουν στο σύντη του Λονδίνου πληρώνουν 7% του εισοδήματό του για την αγορά τροφίμων. Στις κομιτείες ε, της Μεθορίου Βουλγαρίας, Ρουμανίας το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 50%. Η τιμή των αυγών πετάχτηκε στα ύψη, στην Ουγγαρία για παράδειγμα. Και αυτό οδήγησε τον κόσμο να είναι κατά των μέτρων προστασίας των ζώων. Διότι οι άνθρωποι στο κάτω της γραφής θέλουν να γεμίσουν το τραπέζι τους. Αυτά θέλω να θυμίσω, διότι αυτά είναι τα πρώτα που πρέπει να μας απασχολήσουν, δηλαδή οι ανησυχίες των καταναλωτών αυτοί που θα πάνε στο κατάστημα και θα διαλέξουν το προϊόν, αυτοί θα κρίνουν εν τέλει. Δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μόνο τις απόψεις οργανωμένων ομάδων οι, οι οποίοι ασκούν πίεση. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να ακούμε τους ε, Χορτοφάγου για τον τρόπο που θα παραχθεί το κρέα διότι αυτή δεν πρόκειται να φάνε ποτέ κρέας. Το σωστό λοιπόν θα ήταν, το σωστό βήμα προς τα εμπρός θα ήταν να ρωτήσουμε τους καταναλωτές, να παρακολουθήσουμε την συμπεριφορά των καταναλωτών, να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτοί καταναλώνουν και τότε να διατυπώσουμε προδιαγραφές των οποίων εφαρμογή να παρακολουθείτε από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εν τέλει, όπως είπα, ο καταναλωτής είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει τελικά τι θα αγοράσει και τι όχι. Και βέβαια η παραγωγή που παράγουν προϊόντα που θα απευθυνθούν σε αγορές όπου οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω, ε, αυτοί βεβαίως θα παραγάγουν έτσι, αλλά οι παραγωγή η οποία διαθέτουν τα προϊόντα τους σε αγορές όπου οι προσδοκίες δεν είναι τόσο υψηλές, ε, τότε αυτή θα είναι ε, ικανοποιημένοι και με λιγότερα. Συχνά ο καταναλωτής δεν γνωρίζει διόλου τι ακριβώς αγοράζει, από που προέρχεται αυτό που αγοράζει. Για παράδειγμα, στα αεροπλάνα, στα αεροπορικά ταξίδια ή σε εστιατόρια. Σας προσφέρετε ένα προϊόν που υποτίθεται ότι είναι, ε, είναι μαγειρεμένο σύμφωνα με τις επεπιθύσεις διαφόρων εκκλησιών, διαφόρων αριθρησκειών κτλ. Ich έχουμε το βασικό πρόβλημα στην προστασία των ζώων, ότι έχουμε διαφορετικές ταχύτητες στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Αυτές οι διαφορετικές ταχύτητες δεν πρόκειται να αλλάξουν στο προσεχέ μέλλον, διότι οι χώρες εκείνες μέλη οι οποίες κατέβαλαν προσπάθεια και κόπο για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις, εκεί οι γεωρικές εκμεταλλεύσεις εν τέλει των χωρών αυτών δηλαδή έχουν το συγκριτικό μειονέκτημα, διότι άλλοι δεν σεβάστηκαν τους ε, κανόνες αυτούς. Άρα για τις προθεσμίες θα πρέπει να γίνει και διάκριση μεταξύ της νομικής εφαρμογής και της πρακτικής εφαρμογής. Δεν είναι δυνατόν χώρε οι οποίε μετέφεραν το νομοθέτημα στην ε, ενωμή τάξη του, αλλά και το εφάρμοσαν στην πράξη, εν τέλει όπω είπα υφίστανται το μειονέκτημα απέναντι σε χώρε, οι οποίε ναι μεν το μετέφεραν στην ενωμή τάξη τους αλλά στην πράξη δεν το εφάρμοσαν. Εκεί χρειάζεται να, δείτε, να δίνονται μεταφατικέ περίοδοι και στι πρώτε χώρε, ώστε να μην υπάρχει μειονέκτημα, ε, συγκριτικό μειονέκτημα ανταγωνιστικότητα. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν λαμβάνουν πολύ υπόψη είναι το κόστος των επενδύσεων που είναι υψηλά και χρειάζονται για παράδειγμα 20 χρόνια απόσβεσης. Εάν λοιπόν κάθε 20 χρόνια ζητούμε αλλαγές και επομένως και νέες επενδύσεις δεν προλαβαίνει ο Γιώργος καν να αποσβέσει την επένδυσή του. Πώς θα εξοικονομήσει για να μπορέσει να προχωρήσει στην επόμενη επένδυση. Ας μην απορούμε λοιπόν που οι αγρότες λένε ότι αυτό, αυτό το κόστος μας καταστρέφει και μην λησμονούμε ότι το κόστος της προστασίας των ζώων είναι ένα μέρος μόνον του κόστος που είναι ε, ε, ε, διατεθειμένος να δεχθεί ο καταναλωτής. Υπάρχουν κόστη και από αλλού και τελικά κάνουν την κατάσταση πολύ δύσκολη. Τώρα για τις διμερείς συμφωνίες. Και εδώ θα πρέπει να παραμείνουμε κάπως ρεαλιστές. Να λάβουμε υπόψη ότι η αύξηση του πληθυσμού ανά τον πλανήτη δεν θα είναι στην Ευρώπη οι αλλαγέ στι αγορέ λοιπόν θα γίνουν, και, θα γίνουν αλλού και αυτοί δεν πρόκειται να δεχτούν από εμάς να τους υπαγορεύσουμε κανόνες προστασίας των ζώων. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ η στάση και η θέση και της αγροτικής οικονομίας να είναι σαφέστερη αλλά και ειλικρινέστερη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω την αγροτική οικονομία από τις διμερείς συμφωνίες. Και δύο λόγια ακόμα για τον καταναλωτή γενικότερα. Ωραία είναι να, θέλουμε να ρωτήσουμε τον καταναλωτή. Όταν ήμουν νεότερη έμαθα ότι αν ρωτήσουμε τον πολίτη τι κάνει, άρα θα μας πει από αυτά που θα κάνει στο τέλος τα ευχολόγια του καταναλωτή είναι τεράστια, όπως τα γράμματα που στέλνουν τα παιδιά στον Άγιο Βασίλη. Στην πραγματικότητα όμως ο καταναλωτής όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ άλλα κάνει από αυτά που έχει δηλώσει προηγουμένως. Σας παρακαλώ, ο επόμενος ομιλητής, ε, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το επόμενο σημείο. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω, το έγγραφο. Το σε μεγάλο βαθμό αλλά νομίζω ότι κάτι λείπει. Σε ορισμένες περιοχές ε, γίνεται μεγάλη κουβέντα για αυτό το θέμα, σε άλλες δεν το συζητάμε καθόλου. Ξέρουμε ότι ας πούμε ε, μερικές φορές ε, ταΐζουμε υπερβολικά πολύ τα ζώα. Ε, παραδείγματος χάρη ε, τις γαλοπούλες φερρυπίν. Τις κάνουμε τόσο παχές που δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος τους. Επίσης, ο χημικός ευνοχισμός των χείρων ή άλλα στοιχεία μεταχείριση των ζώων. Δεν τα αναφέρουμε στο κείμενό μα. Δεν τα λέμε ξεκάθαρα όλα αυτά. Πρέπει να πούμε ποια είναι η πολιτική που υποστηρίζουμε. Ή να πούμε ότι δεν θέλουμε καθόλου τέτοιου τύπου πολιτικές. Eh, Ευχαριστώ. Λοιπόν, λυπούμε που δεν ήμουν παρούσα από την αρχή της συζητήσεως. Ήμουν όμως σε άλλη συνεδρίαση. Η προστασία των ζώων είναι πολύ σημαντική από γενικότερη άποψη. Ας μην αντιπαραθέτουμε τις δύο πλευρέ από τη μια μεριά του αγρότες και από την άλλη μεριά τα συμφέροντα των ζώων. Αυτό που είδα εγώ είναι ότι για τον καλό αγρότη Πάντοτε είναι σημαντικό το ζώο να είναι σε καλή υγεία και σε καλή κατάσταση. Και αυτή η καλή διαβίωση των ζώων σημαίνει και κατάλληλη εκτροφή τους. Και το καλύτερο είναι να γίνεται σε μικρές εκμεταλλεύσεις, σε πολυλειτουργικές ε, εκμεταλλεύσεις. Όπου εκεί σημειώνονται και τα λιγότερα προβλήματα σχετικά με την διαβίωση των ζώων. Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας τροφίμων, η δημιουργία ε, θέσεων απασχόλησης, αυτή επίσης εξασφαλίζεται σε αυτές τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι αυτές οι μικρές εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο λόγω του ευρωπαϊκού φαινομένου αρπαγής της γης, δηλαδή κερδοσκοπίας κερδοσκοπικής αγοράς γεών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει και αυτό το πρόβλημα. Είναι εν τέλει δική μας ευθύνη να αντιμετωπιστούν οι κερδοσκοπικές αυτές τάσεις. Γίνονται κερδοσκοπικές αγορές γης στην Ουγγαρία που οδηγούν σε σημαντική, σε δημιουργική θέση της εκμεταλλεύσης, της αγροτικής εκμεταλλεύσης. Ας μην εισμονούμε ότι και αυτό αποτελεί ένα τμήμα του συνόλου. Θέλω λοιπόν η Επιτροπή Γεωργίας να εξετάσει και αυτό το λεγόμενο στα αγγλικά land grabbing. Ευχαριστώ να απαντήσει κυρία Πόλσεν. Ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις. Επαναλαμβάνω, ακόμα μία φορά, ο στόχος μου είναι να καταλήξουμε σε μια απλή, σαφή και χρήσιμη νομοθεσία. Σήμερα τα νομοθετήματα είναι πολύ τεχνικά, πολύ μπερδεμένα, πολύ εκτεταμένα. Δεν μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα καταλάβουν. Ίσως γίνω λίγο δυσάρεστη τώρα, τώρα στο τέλος. Αν θέλετε να συμμετάσχετε στην απλούστευση και στη διευκρίνηση της νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων, μην παρουσιάστε πολύ περίπλοκες τροπολογίες. Σας παρακαλώ να είσαστε απλοί. Σας ευχαριστώ πολύ την εισηγήτριά μας. Ευχαριστώ κυρία Μάριτ Πόλσεν. Αν δεν θέλει κανένα άλλο το λόγο, νομίζω ότι έχει ε, ολοκληρωθεί η συζήτηση σε επίπεδο επιτροπής. Θα τα πούμε αύριο στις 10 και τώρα να παραμείνουν οι συντονιστές. Α, όχι, διορθώνει ο Πρόεδρος. Αύριο θα, συζητήσει, θα συνέλθει η Επιτροπή μας στις 9.30, όχι στις 10. Οι συντονιστές θέλουν να παραμείνουν, γιατί έχω μια συνάντηση με τους εκπροσώπους της συνέλευση των πολιτικών χωρών. Θα ήθελα οι συντονιστές των ομάδων να παραμείνουν λοιπόν στην αίθουσα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι να εξέλθουν. Θα τα ξαναπούμε όλοι μας αύριο στις 9.30. Αύριο το πρωί στις 9 θα συνεδριάσουν ξανά οι συντονιστές και στις 9.30 ε, θα συνεδριάσει η Επιτροπή. Θα ήθελα οι συντονιστές να καθίσουν παρακαλώ για να αρχίσει η συνεδρίαση.